Οπότε θα δοθεί ευκαιρία τώρα στον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμαν να καθίσει και η κυρία Γκάλπελτς θα αναλάβει την Προεδρία της Συνόδου. Αξιότιμα μέλη, ε, συνεχίζουμε λοιπόν. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ε, τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Τίμερμαντς. Πρόεδρε, τους τελευταίους έξι μήνες ε, αν προηγουμένου ε, αριθμός ανθρώπων έφτασε στα σύνορά μας και οι μεταναστευτικές ροές αυτές ε, στο προσεχές μέλλον δεν πρόκειται να αντιστραφούν. Δεκάδες χιλιάδες ε, ανθρώπων φεύγουν για να γλιτώσουν από ε, τον πόλεμο. Και η Ευρώπη παραμένει ελκυστική για εκείνους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Ως Ευρωπαίοι δεν μπορούμε ούτε πρόκειται να ε, γυρίσουμε την πλάτη στις ηθικές και διεθνείς νομικές μας υποχρεώσεις να δώσουμε προστασία και εκείνους που τη χρειάζονται. Αλλά δεν μπορούμε ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να έχουμε ανεξέλεγκτες ροές μεταναστών που περνούν γρήγορα προς το βορρά, το ένα σύνορο μετά το άλλο και αυτό έρχεται σε βαθιά και ριζική ε, αντίφαση με τους κανόνες του Σέγγεν και το σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φάνηκαν σοβαρές αδυναμίες από την κρίση ε, σε τμήματα των εξωτερικών συνόρων μας. Αυτό και μια πολιτική τροχονόμου που ακολούθησαν κάποια κράτη-μέλη οδήγησαν ε, σε προσωρινούς ελέγχους στα σύνορα σε κάποιες χώρες, το οποίο θέτει ένα αμφιβόλο το Σέγγεν, το σύστημα και τις ε, ωφέλειες που έχει για τους πολίτες και την οικονομία. 5 με 18 δισεκατομμύρια ετησίως θα μας κοστίσει η κατάργηση του Σέγγεν. Οπότε θα πρέπει να τακτοποιήσουμε τα συστήματά μας και να μπορούμε με αποτελεσματικότητα να αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση Όλο αυτού του κόσμου που ε, είναι στην ε, Φυγή. Άρα χρειάζεται καλύτερη διαχείριση για εκείνους που χρειάζονται προστασία και ταχεία ταυτοποίηση και επιστροφή εκείνων που δεν δικαιούνται να βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στις 10 Φεβρουαρίου ε, παρουσιάσαμε κάποιους στόχου που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την περασμένη εβδομάδα σε συνέχεια αυτών ε, ε, πρόσθεσε ένα οδικό χάρτη για να επανέλθει στην ομαλότητα η ζώνη Σέγγεν μέχρι τα τέλη του έτους. Χαίρομαι που ο οδικός αυτός χάρτης ε, βρίσκει την πλήρη έγκριση των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων όπως διαπιστώθηκε χθε. Στον οδικό μας χάρτη λοιπόν εντοπίζουμε τρεις βασικές προτεραιότητες. Πρώτη, η Ελλάδα χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις σοβαρές δυναμίες που έχει στη διαχείριση των συνόρων με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τους οργανισμούς ε, της Ένωσης και άλλα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμφωνήσουμε σίγουρα και σύντομα για την Ευρωπαϊκή Σύνοροφυλακή και Ακτοφυλακή για να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τα εξωτερικά μα σύνορα και προσβλέπω στο Κοινοβούλιο για να διαδραματίσει το ρόλο που του αναλογεί. Δεύτερη προτεραιότητα. Η ε, προσέγγιση τροχονόμου θα πρέπει να σταματήσει τώρα ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα ε, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση εκείνων που βρίσκονται στην επικράτειά της. Συνεργαζόμαστε στενά με τις ε, ελληνικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς για να αυξήσουμε τη δυνατότητα υποδοχής. Επίσης προτείνουμε ε, ένα νέο μέσο ανθρωπιστικής υποστήριξης Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουμε καλύτερα και ταχύτερα για να ληφθούν οι αποφάσεις ε, για την μετακατάσταση και επανεγκατάσταση και να ε, χαλαρώσει η πίεση που υφίσταται η Ελλάδα. Χαίρομαι που επιταχύνεται τις τελευταίες μέρες ο ρυθμός επανεγκατάστασης. Τρίτον, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες Σέγγεν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ε, την επιβίωση του Σέγγεν. Ο δικός χάρτης δείχνει ότι αν χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση ε, μέχρι το Μάιο ε, για προσωρινούς ελέγχους ως τότε, σε μέρη τμήματα των συνόρων όπου αυτή είναι απαραίτητη και θα είναι περιορισμένη σε χρόνο με σταδιακή κατάργησή του στο Δεκέμβριο θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Ο στόχο δεν είναι να τιμωρηθεί καμία χώρα μέλο. Ε, θα πρέπει να είναι συντονισμένη η προσέγγιση, θα συνεργαζόμαστε όλοι με τρόπο ε, συντεταγμένο μέχρι να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Ε, σε αυτή την κρίση τα πάντα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και θα πρέπει όλα να γίνονται παράλληλα. Καταρχάς θα πρέπει να μειωθούν οι αφήξεις στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό είναι εκ των όνου κάνευ να συνεχίσουμε την συνεργασία μας με την Τουρκία για να εφαρμοστεί πλήρως το κοινό πρόγραμμα ε, δράσης, να σπάσει το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών και να μην χάνονται ζωές και ο μόνος βιώσιμος τρόπος να φτάνει κανείς στην Ευρώπη είναι η νόμιμη διαβλή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να συνεργαστεί και να υποστηρίξει τις επόμενες μέρες ε, με βάση τις αρχές ε, της χθεσινής δήλωσης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Όπως συμφώνησαν οι ηγέτες, ε, θα πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστός ο ευρωπαϊκός και ο διεθνής νόμος. Ταυτόχρονα θα πρέπει η Ελλάδα να επιστρέψει στο σύστημα του Δουβλίνου σύμφωνα με τι συστάσει που κάναμε στι 10 Φεβρουαρίου. Πιο μακροπρόθεσμα θα πρέπει να ε, ξανακοιτάξουμε τον κανονισμό Δουβλίνου έτσι ώστε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου βιώσιμο. Και ένα τελευταίο, χωρίς να είναι αυτό το λιγότερο σημαντικό, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλίσουμε ε, ασφαλείς ε, εναλλακτικές διόδους για εκείνους που χρειάζονται προστασία, για να προστατεύονται εγγυημένα οι ευάλωτοι, μεταξύ αυτών γυναίκες και ανήλικοι. Θα πρέπει και όπως τονίστε και στην ε, σημερινή συζήτηση το πρωί να σκεφτούμε και τις γυναίκες πρόσφυγες και θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που ακριβώς την 8η Μαρτίου έθεσε αυτό το ζήτημα. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε όλα αυτά τα μέτωπα και να τηρούμε τα συμφωνηθέντα. Σε αυτό δεσμεύτηκαν οι ηγέτες σε διαδοχικές συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα θα ήρθε η ώρα των αποτελεσμάτων. Έχουμε σχέδιο και θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αργά αλλά σταθερά το σχέδιο αυτό αρχίζει να υλοποιείται και να αποδίδει καρπούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για τις αρχικές σας ε, αυτές σκέψεις και την ανακοίνωση. Ακολουθούν ομιλητές ε, από τις πολιτικές ομάδες. Πρώτη η κυρία Χόλμαια από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κύριε Αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Καταρχά, θέλω να σα ευχαριστήσω ειλικρινά για την επισκόπηση αυτή, κύριε Τίμερμαν. Ε, είναι γεγονό ότι με μικρά βήματα μπορούμε να προχωρούμε, αλλά δυστυχώ τα βήματα παρά είναι μικρά ακόμα. Γιατί ε, δεδομένου και του μεγέθου χρειάζεται άλλη προσέγγιση για να προχωρήσουμε ουσιαστικά. Τα στοιχεία καταχώρησης σε ποσοστά στην Ελλάδα δίνονται ε, είναι γεγονός αυτό, έχουν αυξηθεί, αλλά πού βασίζονται αυτά τα ποσοστά, γιατί οι πραγματικοί αριθμοί ε, δεν είναι σαφείς, γιατί δεν ξέρουμε καν, το είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν ξέρουμε καν πόσοι συγκεκριμένα περνούν τα σύνορα. Χαίρομαι που στη Σύνοδο Κορυφής με την Τουρκία κάναμε ένα βήμα πρόοδο για συνεργασία με την Τουρκία και περιμένουμε και άλλα βήματα μέχρι τα μέσα του μηνός και θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική από κάποια κράτη-μέλη αφού είναι απλώς να περνούν από το έδαφος τους οι πρόσφυγες. Και θα πρέπει να δούμε πιο πολύ το θέμα της διακίνησης των προσώπων. Το βλέπω στην Ευρωπόλ αλλά και στη Frontex. Έχουν το προσωπικό τους, το οποίο δεν επαρκεί όμως. Και ούτε η ΆΣΟ ούτε η Frontex έχουν στελεχωθεί πλήρως διότι τα κράτη-μέλη δεν αποσπούν τους ε, απαραίτητους εμπειρογνώμονες. Με αυτά τα πράγματα είναι αξιοθενήνητα. Κανονικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, συνεργάζεται τα κράτη-μέλη. Και θέλω να σας παρακαλέσω για το εξή. Το 2014 ήταν 4.000 τα παιδιά που είχαν βαριές κακοποιήσεις σεξουαλικές. Το 2015 ήταν 8.000. Το 2016 μόνο το Γενάρη είναι πάνω ε, από το 2015 τα παιδιά αυτά, τα προσφυγόπουλα, έχουν πέσει στα νύχια των διακινητών και των εγκληματιών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντά σε αυτό και χρειάζεται περισσότερο προσωπικό για να διαχειρίζεται αυτά τα πράγματα και να προστατεύει καλύτερα αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα ε, να σας πω ότι υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην Ουγγρική καμπίνα με τη διερμηνία. Ελπίζω οι τεχνικέ υπηρεσίε να το λύσουν. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σίπελ, εξ ονόματο Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ. Περί τίνος πρόκειται, για ποιο πράγμα συζητούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εφαρμόσει και πάλι το Δουβλίνο στην Ελλάδα. Ένα σύστημα που ουδέποτε λειτουργήσε και που ρίχνει όλη την ευθύνη για τους ε, πρόσφυγες σε χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα. Εάν κλείσει η Βαλκανική οδός, τότε ή αν παραμείνει κλειστή, για να το πω καλύτερα, τότε η κατάσταση στην Ελλάδα ε, οριστικά θα γίνει ανθρωπιστική καταστροφή. Οπότε ποιο Δουβλίνο. Τα άλλα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους. Ανταυτού τώρα φέραμε την Τουρκία να μας λύσει τα προβλήματα και να τα αναλάβει εκείνη. Μα η Τουρκία είναι ασφαλές κράτος και είναι και αξιόπιστος εταίρος. Η νευτική διαδικασία με τους Κούρδους έχει ε, τερματιστεί. Ε, οι δικηγόροι και οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να δουλέψουν. Κάνει κατάληψη σε κανάλια και μετά την Κίνα έχει τους περισσότερους δημοσιογράφους στη φυλακή. Και ερχόμαστε να την επιβραβεύσουμε για τρία εκατομμύρια πρόσφυγες σχεδόν και ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι εμείς ως Ήπειρος με 500 εκατομμύρια κατοίκους ε, είμαστε λέει ιδιαίτερα επιβαρημένοι με τέτοιο αριθμό. Αυτά τα πράγματα είναι αξιοθρύνητα. Χάνει την ε, αξία της η Ευρώπη όχι μόνο ως τόπος σχετικής ευημερίας αλλά και ως τόπος ελευθερίας, δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα αυτό πλήττει τους πρόσφυγες, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μοιραίο μήνυμα που στέλνουμε στους ίδιους πολίτες μας, άνδρες και γυναίκες. Επιτροπή και Συμβούλιο επιτέλους θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους να επιδείξουν ηγεσία και να προχωρήσουν το θέμα του καταμερισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, η καταπολέμηση των αιτίων ε, χρειάζεται καταπολέμηση των διακινητών, η βελτίωση των συνθήκων διαβίωση των προσφύγων στις τρίτες χώρες, όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά μόνο αν αναλάβει ο καθένα τις ευθύνε του θα έχουμε μια πιο ισχυρή διαπραγματευτική θέση και εμεί θα είμαστε από την πλευρά μας αξιόπιστος εταίρο, τον οποίο κανεί μπορεί να υπολογίζει. Έχετε μπλε κάρτα του κυρίου Γιάκοφσιτ, κυρία Ζίπελ. Τη δέχεστε? Yes. Yes. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστώ καταρχήν συνάδελφοι που δεχτήκατε την κάρτα μου. Αναφερθήκατε στο διάδρομο των Δυτικών Βαλκανίων και είπατε πως δεν θα πρέπει να κλείσει. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Η οδός των Δυτικών Βαλκανίων θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Αλλά συμφωνείτε μαζί μου πως θα πρέπει να ξέρουμε ποιος περνάει από αυτή την οδό η Ελλάδα σίγουρα δεν μπορεί να ξαναγκαταστήσει το σύστημα του Δοβλίνου γιατί κατέρευσε εδώ και καιρό. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ποιος μπαίνει στην Ευρώπη, συμφωνείτε μαζί μου. Συμφωνώ ότι η καταχώρηση όλων των αφήξεων θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο. Το είπε και η κυρία Χολμάγερ προηγουμένως. Αυτό δεν μπορεί να βαραίνει μόνο την Ελλάδα, για παράδειγμα, αλλά χρειάζεται υποστήριξη από προσωπικό, από όλα τα κράτη-μέλη. Και αν το καταφέρουμε αυτό και το εξασφαλίσουμε, θα έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κύρκο, που είναι ο επόμενος ομιλητής, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Είμαστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε την εφαρμογή των κανόνων δεν είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, αλλά τελικά οι κανόνες θα μας σώσουν. Γιατί αν δεν παίζει κανείς το παιχνίδι σύμφωνα με τους κανόνες, τότε έχει πρόβλημα. Οι κανόνες και η εφαρμογή δεν επιτρέπουν να κάνει κανείς ε, ανακοινώσεις, να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων κτλ. Αλλά ακούσαμε για δεύτερη φορά από την Τουρκία δεύτερη φορά μέσα σε 12 μήνες πώς τους κανόνες μας τους πετούν στα σκουπίδια. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει στους κανόνες να δώσουμε την ευκαιρία να χρησιμεύσουν. Και δεν θα πρέπει να χαράσουμε νέες πολιτικοί φασιζόμενοι στην απελπισία. Βεβαίως και με πολλές προτάσεις της Κομισιόν συμφωνώ. Και θα πρέπει να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε. Αλλά να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα, να είναι πιο αποτελεσματικές οι επιστροφές, να δείξουμε αλληλεγγύη μέσω της ε, ΆΣΟ και μας είπε ότι πρόεδρος κ. στήμεραν σήμερα ότι αυτά θα συμβούν. Πουθενά όμως ε, στους ήδη υπαγιωμένους κανόνες δεν λέει πως θα πρέπει να αναλάβουμε δράση που θα είναι αντίθετη με τους δικούς μας κανόνες ασύλου να ε, εγκαταλείψουμε τα κριτήρια της Κοπενχάγης και να ξοδέψουμε δισεκατομμύρια για απλές υποσχέσεις. Ναι, η επανεγκατάσταση ακόμα δεν λειτουργεί και φοβάμαι πως οποιαδήποτε συμφωνία γίνει με την Τουρκία, αν δεν υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και αν δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες αναφοράς και ε, δεσμεύσεις δεν θα πετύχει. δεν θα πετύχει σε μια εποχή που χρειαζόμαστε επιτυχίες. Και ο Τζορτ Μπέρναρτ Σό δυστυχώς είχε δίκιο όταν είπε πως Μαθαίνουμε από την ιστορία, αλλά δεν μαθαίνουμε, δεν διδασκόμαστε από την ιστορία. Ευχαριστώ που δέχεστε την μπλε κάρτα. Δεν συμφωνείτε μαζί μου πως η κατάσταση με τη μετανάστευση είναι ο μεγαλύτερος ε, ο μεγαλύτερος παράγοντας για τον οποίο έχει χάσει την επαφή η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους πολίτες και γιατί υπάρχει τέτοια αρνητική στάση από τους πολίτες. Συμφωνείτε μαζί μας πως τα αποπληπισμένα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την κρίση είναι να παρακαλά την Τουρκία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και αυτό αποδεικνύει το πόσο αδύναμοι είμαστε. Ευχαριστώ για τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τις οποίες θα πρέπει να σκεφτώ για κάποιο χρόνο. Αλλά εντωμεταξύ να σας πω το εξής. Αν είχατε ακούσει αυτά που είπα στη δική μου ε, ομιλία, θα καταλαβαίνατε πως αυτό που προτείνω είναι ένας θετικός τρόπος να προχωρήσουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει για να γίνονται και αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο λογικές. Γιατί αν εγκαταλείψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω πως εσείς συνάδελφοι θα το επιθυμούσατε, δεν θα μπορούμε να επηρεάσουμε προς το θετικότερο τις αποφάσεις γιατί ξέρετε πως εγώ είμαι πρώην Υπουργός Μετανάστευσης. Μπορώ να βοηθήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει μια κρίση η οποία είναι απαραίτητο να λυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σεσίλια Βίξτρομ έχει το λόγο από φίλου ελευθέρους Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ήπειρος αντιμετωπίζει έναν αριθμό προσφύγων που φεύγουν από τον πόλεμο χωρίς προηγούμενο και η ανταπόκριση των ηγετών ήταν μάλλον ε, θλιβερή οπότε αυτό που θα πρέπει να γίνει τι είναι συστηματική επαναπρόθεση στα σύνορά μας αυτό είναι ενάντια σε κάθε συνθήκη και σε κάθε δίκαιο είδαμε ότι έχουν ξαναρχίσει έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα και το Μπερτέ μας λέει ότι μόνο το οικονομικό κόστος της καταρρεύσης του Σέγκερ θα είναι 1,5 ε, ε, περίπου 3 ευρώ για οπότε θα, τώρα βλέπουμε ότι συναγωνίζεται το ένα κράτος, το άλλο πιο θα είναι χειρότερο ε, για να αποθήσει τους ε, πρόσφυγες, τους μετανάστες. Αυτό όμως που λείπει είναι ε, μια στιβαρή ηγεσία. Μια στιβαρή ηγεσία για την μοναδική λύση που μπορεί να μας κάνει να ελέγξουμε την ε, κατάσταση. Δηλαδή αυτό το οποίο χρειάζεται είναι κοινή δράση, κοινοτική μέθοδος και έτσι να είναι ε, λογική κατανομή των ευθυνών και αυτό το οποίο έγινε κυρία είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κοινή διαχείριση η υποδοχή κοινή των ε, προσφύγων και επαναπρόθεση αυτών που δεν πληρούν τα διεθνή κριτήρια για προστασία και όλα αυτά να γίνονται με τρόπο αξιοπρεπή. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Τιμερός θα πρέπει να συνεχίσουν τις αξιέπαινες προσπάθειές τους και να κατεβάσουν κάποια πρόταση αυθεντικά ευρωπαϊκή και κυρίως ε, να υπάρξει μεταρρύνση της συνθήκης του Δουρλίνου ήρθε η ώρα να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο και εσεί Επιτροπή και εμεί το Κοινοβούλιο και να εμπλακούν την προσπάθεια οι λίγοι ηγέτε που ακόμη μετράνε. Είναι κάτι το οποίο το αξίζει σήμερα η Ευρώπη. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η Κορνίλια για 1,5 λεπτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ αυτό που βλέπουμε σήμερα να γίνεται με τους πρόσφυγες δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παρακινησμός, διότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πρόθυμα να υποδεχτούν πρόσφυγες και το έχουμε κάνει τώρα ανατολίτικο παζάρι. Δηλαδή θα μου δώσεις ένα παράνομο μετανάστη ε, για να σου δώσω εγώ ένα νόμιμο ε, πρόσφυγα, όπως λέγεται. Έτσι λέει η Τουρκία. Ε, η επαναπροώθηση, η απόθεση των προσφύγων προς την Τουρκία Κατά τα άλλα είναι κάτι το αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο, γιατί μέχρι σήμερα η Τουρκία ε, έχει υπογράψει τη σύμβαση για τους πρόσφυγες μόνο με περιφερειακές επιφυλάξεις. Έχει αποτύχει η ατζέντα της μετανάστευσης, έχει γίνει ατζέντα της καταστολής. Και τώρα εάν κάθεστε και σκέφτεστε να δίνετε προστασία μόνο σε σύρους, και μάλιστα και γίνεται λόγος και για ασφαλείς ζώνες και περιοχές στην Συρία. Ε, είναι ελεηνό αυτό και έχει καταντήσει φάρσα. Και επίσης ε, μας ε, χειρίζεται η Τουρκία που ε, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, καταστέλει τον τύπο και πυροβολεί το λαό της. Το δικαίωμα στο άσυλο είναι ατομικό. Η σύμβαση της Γενέβης καταργείται και μετά το δεύτερο ο παγκόσμιο πόλεμο είναι θέμα πολιτισμού. Εμείς ως αριστερά δεν πρόκειται να το δεχθούμε και δεν θα αφήσουμε μέσων ε, που ε, έχουμε στη διάθεσή μας ως ευρωβουλευτές να κινητοποιήσουμε και την κοινωνία των πολιτών ενάντια σε αυτό. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σαρχεντίνη από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Τίμερμας, κύριε Βραμόπουλε, αυτή ήταν η ευκαιρία που θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας εξηγήσει και εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς τι πιστεύετε για τα χτεσινά συμπεράσματα του Συμβουλίου. Εγώ σας ακούω και βλέπω ε, ε, να λέτε κάτι για πιστή συνεργασία αλλά και ένα disclaimer εντός του νόμου και εντός των διεθνών συνθήκων αλλά ε, βεβαίως θα συνεργαστούμε πιστά με την πρόταση του Συμβουλίου που δεν έχει σκοπό να δώσει εστίες και υποδοχή στους πρόσφυγες αλλά έχει κύριο στόχο να σταματήσει ή να περιορίσει τις εισρωές στην Ευρώπη και από την αρχή, από την πρώτη ε, φάση της ανάλυσης μας, ε, δεν έχουμε καταλάβει ότι οι πρόσφυγες από κάπου φεύγουν για να ξεφύγουν και δεν θα πρέπει κάπου να τους στείλει, αλλά θα πρέπει να τους ε, εντάξεις και να τους προστατεύσεις. Και αυτό δεν γίνεται όταν λες ότι σου δίνω ένα μεταχειρισμένο πρόσφυγα, δώσ' μου ένα φρέσκο καινούριο που έχεις εσύ. Αυτά δεν είναι ε, μεταχειρισμένες φιάλες που τις γυρνάς πίσω και παίρνεις το αντίτιμο. Είναι άνθρωποι που χρειάζονται προστασία. Ποιο θα είναι το νόμιμο λοιπόν και η νόμιμη οδός και πώς θα διοργανωθεί. Και όταν μιλάμε για ελέγχου στα σύνορα θα πρέπει να συζητάμε ε, και για το γεγονός ότι έρχονται παράνομα γιατί δεν μπορούν να περάσουν με νόμιμο τρόπο τα σύνορα. Και τώρα λέτε ε, ελέγχου στα σύνορα. Πρόβλημα ηγεσία και έλλειμμα ηγεσία δεν έχει μόνο το Συμβούλιο αλλά και εσεί. Και είναι κρίμα γιατί ήσασταν σε καλό δρόμο. Η κυρία Φεράρα. Δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και σήμερα ε, μιλούμε και για αυτό το θέμα, για βήματα σημειωτών που κάνουμε. Αυτό όσον αφορά το θεματολόγιο της μετανάστευσης. Μιλούμε για 10.000 ανηλίκους που έχουν εξαφανιστεί. Ε, δεν συνοδεύονται, δεν συνοδεύοντουσαν ουτε τη τότε στην Ευρώπη και είπαμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δίκτυα για τις μαφίες δεν μπορούμε να τα σπάσουμε, να τα διαλύσουμε και βέβαια είναι πάρα πολύ ε, θεωρητικό ότι γίνονται προσπάθειες από την Europol και αποδίδονται κάποια αποτελέσματα από αυτές τις επιχειρήσεις Europol. Είπαμε για τη συμφωνία με την Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε την μεταναστευτική κρίση, αλλά δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε ενώπιον του εκβιασμού. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις ροές από την Τουρκία. Τι είναι, είναι ασφαλής χώρα, όχι. Υπάρχουν εγγύσει δικαιωμάτων εκεί. Όχι. Άρα τι θα γίνει. Θέλουμε να πιστούμε ε, ότι είναι. Υπάρχει ένας δισταγμός να καταλάβουμε τι είναι αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Κάποια κράτη-μέλη αρνούνται την αλληλέγγυα προσπάθεια ε, υποδοχής αυτών των ε, ροών. Αν δεν συνεργαστούν τα κράτη-μέλη δεν θα υπάρξει τίποτα. Έχετε κάποια ερώτηση. Τη δέχεστε κύριε Βάτμαντς. Κύριε Βάτμαντς. Ευχαριστώ. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι μιλάτε και για τα 10.000 ε, αγνοούμενα παιδιά ανηλίκους. Πάνω από 40 μέλη των φιλελευθέρων την περασμένη εβδομάδα κάναμε ερώτηση σχετικά και ζητήσαμε να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, Πρόεδρε. Και θέλω να ρωτήσω, η δικιά σας ομάδα τι θα κάνει για να βρεθούν τα παιδιά αυτά. Συζητώ με τη Europol και τη Europe for Missing Children θα πρέπει το 2016 να μην επιτρέπουμε τέτοια πράγματα. Έχουν χαθεί 10.000 παιδιά. Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Οπωσδήποτε. Η πολιτική μας ομάδα έχει δεσμευτεί για την υπόθεση αυτών των μη συνδεδεμένων ανηλίκων και έχουμε βάλει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό που θέλουμε να υπάρξει ένα μείζον πρόγραμμα προστασίας για αυτή την τόσο ευάλωτη κατηγορία. Είναι παράδεκτο αυτό που έγινε γιατί ακόμα σήμερα έχουμε χιλιάδες μη συνοδευομένων ανήλικων που εξαφανίζονται χωρίς ε, να υπάρχει κανένα είδος πλέγμα προστασίας. Οπωσδήποτε και εμείς δεσμευόμαστε για αυτό το θέμα. Η κυρία Μαϊέρα έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, τι φάνηκε από αυτή την κρίση του ασύλου που την έχουμε φτιάξει μόνοι μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δράσει εκατοντάδες χελίδες προτάσεις αλλά δεν μειώθηκε ο αριθμός, ούτε ένας λιγότερος δεν ήρθε. Εχθές οι ηγέτες με την κυρία Μέρκελ ε, να πρωτοστατεί ε, έδωσαν στα χέρια του Τούρκου δικτάτορα Ερντογάν την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αξιοθρύνητα αυτά και ικτρά και ε, κάνει εκβιασμούς η Τουρκία και εμείς κάνουμε τεμενάδες στην Τουρκία. Θέλει ε, να μπει πιο γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι ζητάει εμείς και άλλους τεμενάδες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εξαρτάται από την αναξιόπιστη Τουρκία και παίζει επικίνδυνο παιχνίδι με την ελευθερία μας. Και όλα αυτά για να σταματήσει το τσουνάμι του ασύλου. Αυτά δεν ήταν ούτε συμφωνίες ούτε διαπραγματεύσεις. Είναι ένα ιστορικό σφάλμα και θα πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί. Καλό τον ίδιο μου το Πρωθυπουργό να δείξει σθένος και πυγμή, κλείστε τα σύνορα της Ολλανδίας των κάτω χωρών, μην τα δίνετε στα χέρια της Τουρκίας για το λόγο μας και για την ελευθερία του. Και επόμενος ομιλητής από τους μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Παπαδάκης, παρακαλώ τόσο ο λεγόμενος οδικός χάρτης για τη σέγγεν όσο και η κοινή δήλωση της χθεσινής συνόδου επιβραβεύουν τον εγκλωβισμό χιλιάδων απελπισμένων προσφύγων και μεταναστών στην ελλάδα θεωρώντας τον αφετηρία και δεδομένο επιβεβαιώνουν ότι τα κλειστά σύνορα και οι έλεγχοι οι απελάσεις μέσα από τη διαλογή δεν είναι πολιτική μόνο της αυστρίας ή των χωρών του βίζεγκραντ αλλά ενιαία πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης κλεισίματος της στρόφιγγα με την υπογραφή και της ελληνικής κυβέρνησης. κόντρα και στη συνθήκη της γενέβης η ευρωπαϊκή ένωση όχι μόνο δεν αναγνωρίζει ως πρόσφυγες τους αφγανούς που είναι θύματα και αυτοί των υπεριαλιστικών πολέμων αλλά τώρα ακόμα και στους σύριους τους βγάζει οικονομικούς μετανάστες προς απέλαση στην τουρκία. όσο για το δουβλίνο επανέρχεται ενισχυμένο μαζί με νέους περιορισμούς στη χορήγηση ασύλου σαν αυτούς που μόλις πέρασε η γερμανία και μεθοδεύουν και άλλα κράτη ενθαρρύνοντας τις φασιστικές ορδές και όλα αυτά με τον νατο χωροφύλακα στο αιγαίο με πρόσχημα το προσφυγικό νομιμοποιώντας τις προκλητικές αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της ελλάδας από την αστική τάξη της τουρκίας ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά του ιμπεριαλιστικού πολέμου που προκαλεί η προσφυγιά. αλληλεγγύη στους πρόσφυγες σημαίνει να μεταφερθούν άμεσα στις χώρες τελικού προορισμού τους σημαίνει προσωρινή χώρη ανθρώπινης αξιοπρεπούς φιλοξενίας αλληλεγγύη σημαίνει ένταση της πάλης ενάντια στην πολιτική καταστολή της ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεων και των κρατών μελών της ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στη μήτρα του το καπιταλιστικό σύστημα. Το λόγο έχει η κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα. Έχετε διαδικαστικό. Ε, κοιτάξτε, έχω ε, παρακαλώ να ζητείτε από τους ομιλητές να μιλούν πιο αργά. Δεν τους προβαίνουν οι διερμηνείς. Παρακαλώ να το ζητάτε από τους ομιλητές να μιλούν πιο αργά για να μπορούν να τους προβαίνουν οι διερμηνείς και να κάνουν τη δουλειά τους. Για να καταλαβαίνουμε ακριβώς. Όσοι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα, πολλέ φορέ δεν καταλαβαίνουν τι λέγουν οι ομιλητέ. Η πρόεδρο. Σα ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Παρακαλούμε οι διερμηνείς να προσπαθούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη, αλλά θα πρέπει και οι συνάδελφοι να επιβραδύνουν το ρυθμό του τόσο ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Και τώρα, τρολόγη κυρία Μετσόλα, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι συνεπής, γιατί ξεκάθαρα έχει δεσμευτεί ούτως ώστε να σημειώσουμε κάποια πρόοδο στην αναχέτηση αυτής της κρίσης και θα πρέπει να έχουμε κάποια ευρωπαϊκά εργαλεία και να γίνει τελικά η εφικτή πιο καλή λύση όσον αφορά το Σέγγεν ε, είναι ακρογωνίας λίθος τη σημερινή Ευρώπη. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει το χέρι μα, ώστε να εξασφαλίσουμε λίθος να μείνει στη θέση του αλλά. Ταυτόχρονα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε στροφή σήμερα στην Ευρώπη. Είναι γιατί οι συμπολίτε μα ε, απέσπασαν την υπόσχεση ότι τα εξωτερικά σύνορα θα είναι ασφαλή και ότι θα ε, υπάρχει πληροφόρηση του ενό ε, από τον άλλο. Επομένω, όλα αυτά σήμερα είναι αλληλένδετα και είναι απαραίτητο το για την ασφάλεια. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και πολιτικά αναγκαίο και οικονομικά. Διαπιστώσαμε ότι αν ξαναστήσουμε ελέγχου στα σύνορα ε, θα έχουμε κάθε χρόνο 5 έως 18 δις ευρώ. Άρα θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των συνόρων και ότι θα πρέπει ακριβώς να είναι σε υψηλό επίπεδο αυτός ο έλεγχος των συνόρων. Οπότε το να έχουμε φυλακή, να έχουμε ακτοφυλακή είναι κάτι απαραίτητο και θα πρέπει αυτό να γίνει και ταυτόχρονα θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα προβλήματα της εθνικής κυριαρχίας, να εξασφαλίσουμε το ότι ε, αυτό το κοινό σχέδιο δράσης με την Τουρκία να εφαρμοστεί και αυτό επίσης ε, και να ληφθεί υπόψη προς τούτο ως τη και χθες το βράδυ ε, θα πρέπει όλοι να λάβουν τι υποχρεώσει του για τα εξωτερικά σύνορα και αυτού και, για την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε τι δυσκολίε που ιδίω η Ελλάδα αντιμετωπίσει. Αλλά όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Είναι αυτή η αρχή που προποθέτει τη δράση προ αυτό το μέτωπο. Και κατακλείδη, Πρόεδρε, νομίζω ότι οι συμπολίτε μα απαιτούν από την Ευρώπη να αναλάβει δράση. Χρειάζονται κατεπίγουσε λύσει στα κατεπήγοντα. Τέτοια προσέγγιση πρέπει να γίνει. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Έχετε μια μπλε κάρτα, μια ερώτηση. Δέχεστε, πρόκειται τον κύριο Σόνι. Από τον κύριο Σόνι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσατε κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μετσόλα. Αργά, αργά, μία ε, απάντηση δώστε μου. Βλέπετε κάποια λύση, κάποια λύση για αυτά τα προβλήματα. Θα μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο ούτως ώστε να πείσουμε την εμπλέκουσα μειοψηφία, δηλαδή εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία διστάζουν και δεν θέλουν να προχωρήσουν χέρι-χέρι με για αυτές τις αποφάσεις. Κυρία Μέτσολα, μπορείτε να απαντήσετε. Παρακαλώ, σιγά σιγά. Δεν μπορούν να σα παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Μητσόλα. Και διότι τώρα, ξέρετε, συντάσσω κάποια έκθεση η οποία τον επόμενο μήνα θα περάσει στην Ολομέλεια. Και ακριβώ εκεί εντοπίζουμε το τι γίνεται, ποιε είναι οι απόψει ε, του ε, Κοινοβουλίου. Ε, μετά από τόσα χρόνια που τα κουβεντιάζουμε, ιδίω αυτό έχει γίνει και σε άλλα θεσμικά όργανα μετά από τόσες κουβέντες τελικά αποδέχθημεν το ότι η μετανάστευση και οι σχετικές προκλήσεις είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουν ε, και οι 28 όλα τα κράτη-μέλη. Επομένως χρειάζεται να υπάρξει κατανομή της ε, ευθύνης σε όλους, έτσι βρεθεί μόνο η Πρόεδρος. Κύριε Μωρά, εσείς το επόμενο έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και ο κύριος Τίμερμαντς, γιατί μας είπε πως έχει κάποιο σχέδιο. Πολλά σχέδια παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά με ακυρεότητα. Και ξέρετε πόσα εκατομμύρια πρόσφατα εστάλθηκαν στην Ελλάδα. Κάτι πολύτιμο λοιπόν μπορεί να συμβεί με το ανθρωπιστικό αυτό εργαλείο, αλλά προφανώς δεν επαρκεί. Και γνωρίζουμε πως πολλά από τα μέλη που ασχολούνται με την κρίση και κάνουν κάτι γνωρίζουν πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και δύο χρόνια τουλάχιστον έχει σχέδια. Το πρόβλημα είναι το Συμβούλιο είναι η επιθετική, για παράδειγμα, πολλές φορές χαόδης αντίδραση σε διάφορα σημεία. Οπότε έχουμε δύο ε, διαφορετικές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, αντιμετωπίζουν το πιο δύσκολο που είναι το Δουβλίνο που πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιους, ε, κάποιες υπηρεσίες για τα σύνορα για παράδειγμα ή ΕΑΣΟ δηλαδή βασικές αναθεωρήσεις που χρειάζονται μήνες και όπου όλοι θα χρειαστεί να δουλέψουμε εδώ ε, σε αυτή την αίθουσα και μετά έχουμε και το σχέδιο για την Τουρκία. Και με τα λίγα δευτερόλεπτα που έχω, θέλω να σας πω πως δεν... Να είμαστε προσεκτικοί με το σχέδιο για την Τουρκία, να προσέξουμε, να μην καταπιτάσουμε το διεθνές δίκαιο, να μην εγκαταλείψουμε τις ιδέες μας. Δεν είναι πολυτέλεια αυτή. Δεν μπορούμε εμείς να μην κάνουμε τη δουλειά μας στο Κοινοβούλιο για κάποια από τα βασικά θέματα με τα οποία θα έρθει αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι ε, δυνατόν να αφήνουμε ανθρώπους να πεθαίνουν ή να τραυματίζονται ή να αφήνουμε ε, νέα συνόδευτα παιδιά να χάνονται. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Γιούρικ, κύριε... Συνάδελφε, ναι, κύριε Γιούρικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Εσεί επικρίνετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όμω πριν από δέκα μήνε ήταν οι ειδικέ μα κυβερνήσει οι οποίε πρότειναν το μοναδικό λογικό μηχανισμό που θα μπορούσε να έχει σταματήσει εκείνη τη στιγμή αυτή την ανθρώπινη τραγωδία. Δηλαδή, είχαμε πει τότε πως χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για να κατοπολεμήσουμε την παράνομη ε, διακίνηση ανθρώπων. Δεν είναι αυτό ένα απαραίτητο στοιχείο έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθούμε τους ανθρώπους χωρίς να μεγενθύνουμε το πρόβλημα. Στο σημείο που να γίνεται δυσεπίλητο. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα για το Συμβούλιο δεν είναι αν θα τους ε, καταγγείλουμε ή όχι σε γενικές γραμμές. Νομίζω το πρόβλημα είναι οι ακρότητες στο Συμβούλιο, γιατί υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία προσπαθούν ε, να ε, αποδεχτούν τι ευθύνε του και άλλοι αποποιούνται των ευθυνών του. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν κάποιε χώρε να κάνουν τα πάντα και κάποιε άλλε χώρε να παρατηρούν αδιάφορα αυτού που κάτι κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχέδια και τα σχέδια αυτά έχουν οριμάσει τα τελευταία δύο χρόνια. Και είμαστε πια σε θέση να δράσουμε. Αλλά δυστυχώ όχι γιατί κάποιοι στο Συμβούλιο ήταν επιθετικά διάφοροι. Ευχαριστώ. Η κυρία Στέβενς έχει το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Στο παρελθόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι κυβερνήσεις δεν έδωσαν αρκετή προσοχή στο θέμα της φύλαξης των συνόρων και γι' αυτό ε, ε, καταντήσαμε να είμαστε εξαρτημένοι από την Τουρκία. Δεν μπορούμε πια να ελέγχουμε μόνοι μας τα ίδια μας τα σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη ευάλωτη για να την εκβιάζει η Τουρκία η οποία το ε, καταχράται αυτό πλήρως και αγρίως. Ε, ε, έχουμε τώρα ακολουθήσει τη γραμμή Μέρκελ και βρισκόμαστε σε αυτή τη δινή κατάσταση. Το κόμμα μου, το NVA, ξέρει τι φταίει. Εν περιπτώσει, τώρα δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος και να καταφέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, μπορεί να διαχειρίζεται μόνη της τη μοίρα της και να μην εξαρτάται από χώρες όπως η Τουρκία. Να κλείσουν οι ε, οδοί προς τη ε, Δυτική Ευρώπη, να υπάρχει μια ισχυρή πολιτική αποθήσεων, pushback στην περιφέρεια και με ποσοστώσεις να ελέγξουμε τις ροές. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Μλίναρ. Ένα λεπτό. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω μια ειλικρινή συζήτηση. Στην ανακοίνωση ακόμα συζητούμε την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στι αποφάσει για τι επανεγκαταστάσει. Μα αυτά δεν δουλεύουν, δεν λειτουργούν. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από μια χώρα όπω είναι η Ελλάδα να κάνει hot spots και να είναι και λειτουργικά εάν δεν υπάρχει καταμερισμό. 536 πρόσωπα από τις 66.400 έχουν επανεγκατασταθεί. Αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είμαι πεπισμένη για τα εξή δύο. Πρώτον, πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε εξωτερική ανάθεση των προβλημάτων μας. Ε, χρειάζεται ε, ευρωπαϊκή λύση για το προσφυγικό. Και δεύτερον, συγκεκριμένα μέτρα με έμπρακτη αλληλεγγύη και επιμερισμό ευθυνών αρχίζοντας από τώρα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανέλθει πλήρως η λειτουργία του Σέγγεν εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αλλά έχω το φόβο ότι αυτό είναι μια ασαφής ε, δέσμευση με πολύ μακρινή ημερομηνία. Αφήστε τα λόγια. Χρειάζεται και νόμιμος τρόπος και ασφαλής να έρχονται στην Ευρώπη. Και περιμένω την πρόταση για την γαλάζια κάρτα, για την νόμιμη οικονομική μετανάστευση. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ε, είχατε ένα λεπτό μόνο. Ε, για την ομιλία αυτή. Το λόγο έχει η κυρία Μόλιν Πιόρκ. Ε, Παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, η Σέγγεν θα πρέπει να ξαναλειτουργήσει, αλλά θα πρέπει και η Ευρώπη αντί να κάνει κάποιες επίγουσες διαδικασίες για να δέχεται προσφυγές, πρόσφυγες με συγχωρείτε, θα πρέπει να προετοιμάσει ένα πρόγραμμα που ε, θα σταματά από τους ανθρώπους αυτούς να σταματάνε να φτάνουν στην Ευρώπη. Αυτό κάποιος πρότεινε και είναι απαράδεκτο γιατί με τον τρόπο αυτό αφήνουμε τη λύση σε μια αυταρχική κυβέρνηση αυτή της Τουρκίας παρόλο που έχουμε το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή ε, στο Αιγαίο δεν νομίζω πως έχουμε επιλέξει την κατάλληλη λύση που θα δώσει αποτελέσματα στο μέλλον. Για το μέλλον χρειαζόμαστε μια κοινή διαχείριση της κρίσης στην Ευρώπη. Μια διαχείριση κατά την οποία η Ευρώπη αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Διαφορετικά είμαστε καταδικασμένοι να βρεθούμε σε μια Ευρώπη που καταραίει και που δεν υπερασπίζεται πια τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στο άσυλο. Ευχαριστώ πολύ. Αφήνω το λόγο στην κυρία Κέλλερ για ένα λεπτό. Από τις 10 ε, Ιανουαρίου μας είπατε ποια είναι η ασφαλής τρίτη χώρα. Από τις 10 Φεβρουαρίου με συγχωρείτε έχουμε κάποιες διασφαλίσεις και εχέγγυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπει με τον τρόπο αυτό να τους καλύπτουμε όλους. Μα είναι αυτό έξυπνο, είναι λογικό. Γιατί τοποθετήσαμε αυτά τα εχέγγυα και τις ε, δικλείδες ασφαλείας. Γιατί έχουμε όλους αυτούς τους νόμους και τους κανόνες αν δεν θέλουμε να τους τηρούμε και μετά να λέμε ότι καλά αυτό είναι άσχετο. Οπότε σας ρωτώ το εξή. Πιστεύετε πως η Τουρκία, μια χώρα η οποία στέλνει στρατιώτες εναντίον του ίδιου της του πληθυσμού. Είναι μια χώρα που στέλνει πρόσφυγες πίσω στη Συρία. Ακούμε πως έχουν ε, σκοτώσει ε, οι συνοριοφύλακες, έχουν πυροβολήσει σύρους πρόσφυγες. Πιστεύετε ότι η χώρα αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί τρίτη ασφαλής χώρα όπως περιγράφεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει η κυρία Βίνμπερκ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Τίμερ μας μας είπε ότι υπάρχουν προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα. Πώς μπορεί κανείς να διαφωνίζει ε, λέμε τώρα ε, για το πώς θα συγκροτηθεί μια σύνορια φυλακή. Τριπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός της ε, Frontex. Πρόκειται νόμιζε για έλεγχο των συνόρων. Μα ε, όπως τα είπατε εσείς, πρόκειται για τις κυρίως αρμοδιότητες που είναι η διάσωση. Επομένως, ε, έχουμε τώρα και την ακτοφυλακή. Υπάρχουν ε, επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, τι θα κάνει η συνοριοφυλακή ή η ακτοφυλακή θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή των προσφύγων. Επίσης μας αναφέρατε για 160.000 προσφύγων που θα κατανεμηθούν. Όμως, τι θα γίνει εάν δεν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερου προσφύγους όταν οι πρόσφυγες όταν οι ποσοστώσει εξαντλήθουν θα αναθεωρηθούν αυτέ οι ποσοστώσει. θα αναθεωρηθεί από το σύστημα κατανομής, διανομή μεταξύ των διαφόρων χωρών μελών. Τι θα γίνει η πρόεδρο. ο κ. Μπρίβα είχε το λόγο για ένα λεπτό Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι 700 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που θέλει να διασπαθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό που θα ονόμαζα τον πίθο των Δαναίδων που είναι η πολιτική υποδοχή των ε, μεταναστών. Ακούγοντας τέτοια αριθμητικά στοιχεία σκέφτομαι τους κατοίκους του Καλέ και της Grand Σεντ που υφίσταται τις άμεσες συνέπειες αυτής της ελεύθερης πολιτικής της μετανάστευσης και τις οικογένειες αυτές σκέφτομαι που δεν μπορούν να ζουν με ασφάλεια ή και τους εμπόρους που βάζουν λουκέτο ή και τις γυναίκες αυτές που ε, όπως στην κολονία έπεσαν θύματα πολλαπλών σεξουαλικών επιθέσεων από μετανάστες που δεν έχουν τον παραμικρό σεβασμό για τους νόμους της χώρας στην οποία φτάνουν. Αντί λοιπόν να χρηματοδοτούμε τέτοιες δαπάνες ε, για την ε, μεταναστευτική επιδρομή θα πρέπει τα λεφτά μας να χρησιμεύουν για να καταστρέφονται οι παράνομοι καταβλισμοί και να επιστρέφουν οι λαθρομετανάστες. Να βοηθήσουμε την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία την Ελλάδα να ε, ασφαλίσουν τα ε, σύνορά τους και να σταματήσουν τις ροές των μεταναστών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκολνής έχει το λόγο. Παρακαλώ το ελάχιστο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση ε, που κατατέθηκε πριν από 20 μήνες είναι και αναποτελεσματικό και μη λειτουργικό και πλήρης αποτυχία. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά όταν το βασικό αυτό του θεματολογίου βασίζεται στην περισσότερο ή λιγότερη καλή βούληση ε, της ε, κυβέρνησης μιας τρίτης χώρας, εμπροκειμένου της Τουρκίας με την οποία χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί σχέσεις αμφίσιμες για να μην πω σχιζοφρενείς. Ε, και μάλιστα το εκμεταλλεύεται αυτό η κυβέρνησή της γιατί έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά πόσο αδύναμη είναι η Ευρώπη που είναι στριμωγμένη στο δόγμα της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων και στην επιθυμία της να υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες ε, μετανάστες παρά την αντίθετη άποψη και την εχθρική των λαών της. Και τώρα έχουμε παζάρια όλο και πιο απαιτητικά. Έχετε δώσει στα χέρια του κυρίου Ερντογάν ένα πυρηνικό όπλο του έχετε αναθέσει να φυλάσει εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχει τη δυνατότητα να ανοίγω κλείνει τη στρόφιγγα της μαζικής μετανάστευσης. Το σύστημα ένας προς έναν που υποστήριξε η κυρία Μέρκελ, δηλαδή που τάζει να δεχτεί η Ευρώπη, ένα νόμιμο πρόσφυγα για κάθε λάθρομετανάστη μετανάστη που πιάνεται ή παναπροωθείται στην Τουρκία δεν είναι απλώς νοσηρό αλλά είναι και καταδικασμένο να αποτύχει. Γιατί τελικός προορισμός των νομίμων προσφύγων δεν έχει λυθεί. Τα περισσότερα κράτη-μέλη αρνούνται να συμμετέχουν στο σύστημά σας ποσοστώσεων επανεγκατάστασης. Και επιπλέον οι διακινητές ε, και βάζω στοίχημα έχουν ήδη σκεφτεί πώς θα το εκμεταλλευτούν και αυτό. Και έλεγε ο Αλβέρτο Άινστάιν ότι δεν αλλάζεις ένα σύστημα με τις ίδιες ιδέες, με εκείνες που το δημιούργησαν. Και νομίζω ότι είχε και δίκιο ο άνθρωπος. Η Πρόεδρος, ε, μπλε κάρτα έχετε από τον κύριο Βιοσλόφσκι, τον δέχεστε. Δέχεστε μια ερώτηση με μπλε κάρτα. Κύριε Γκολνής, έχετε ερώτηση με μπλε κάρτα, τη δέχεστε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι η συμφωνία με την Τουρκία είναι απαράδεκτη. Οφελεί κατά παράδεκτο, σκανδαλιστικό τρόπο την ε, Τουρκία. Εξεβιάστησαν οι δημοκράτες των Βρυξελών από τη χώρα αυτή. Ε, με τη σύναψη αυτής της συμφωνίας να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορεί να έχει ασφαλή εξωτερικά σύνορα. Ανέθεσε την ασφάλεια των σύνορων στην Τουρκία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γκολνίσου. Μάλιστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα παζάρι απαράδεκτο και έτσι ε, παροξύνονται οι μεταναστευτικές ε, ρωσιδίες με την κατάρριξη της βίζας και έχουμε επίσης και μετανάστευση από την ίδια την Τουρκία. Ε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που θέλουν να μεταναστεύσουν με ε, προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πρόεδρος. Κύριε Τζαμπόφσκι. Συγγνώμη που δεν προφέρασα το όνομά τη. Αλλά τελικά καταλάβω τι ήθελα να πω. Ο επόμενο τώρα, ο κύριο Μπρόγκ το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις του περασμένου ε, μηνός και της περασμένης εβδομάδες. Διατήρησε την ψυχραιμία της σε μια ε, ε, κατάσταση που κανείς δεν περιμένει. Εδώ προέρχεται για μετακινήσεις ε, μαζικές λαών και θα πρέπει να διατηρηθεί και να σωθεί το Σέγγεν και να διατηρηθεί η κατάργηση των συνοριακών ελέγχων με οδικό χάρτη έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την πηγή της ευημερία μας και των κοινωνικών συστημάτων που είναι εσωτερική αγορά και να μην πληγεί. Θα πρέπει να επανέλθει η εσωτερική τάξη η Σύμβαση της Γενέβης συνάδει και με την εσωτερική τάξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αντιφατικά. Σήμερα αυτό δεν το καταφέρνουμε, αλλά μπορούμε αυτούς τους δύο στόχους να τους επιδιώκουμε από κοινού. Και αυτή είναι πάγια επιθυμία και αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα γίνεται λόγος για συνοριαφυλακή και για ακτοφυλακή ευρωπαϊκή και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι 15 χρόνια, 20 χρόνια Σέγγεν ε, ε, και Δουβλίνο, οι Γερμανοί ε, κάπως την έχουν βγάλει φθηνά και τα έχουμε αφήσει όλα στη Μάλτα, στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Θα πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας για να προχωρήσουμε ο καθένας με τακτοποιημένο τρόπο και διαδικασίες με τους, για τους πρόσφυγες και χρειάζεται εκεί βοήθεια της Τουρκίας. εκεί που βρίσκονται οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν ε, ανθρώπινες συνθήκες για να ζουν και νομίζω ότι το Συμβούλιο τα έχει υπόψη όλα αυτά και θα τα συνεχίσει την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάιντεν Χελτσέρ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο. η σημερινή κρίση πώς προέκυψε μεταξύ άλλων, διότι τα ευρωπαϊκά εργαλεία και μέσα που έχουμε δεν λειτουργούν. Γιατί δεν έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευση με το Δουβλίνο, το οποίο Δουβλίνο επίση δεν λειτουργήσε ποτέ. Είναι θετικό τώρα που έχουμε ένα συνολικό πακέτο με νομοθετική δέσμη μέτρων που θα πρέπει να συζητήσουμε και είμαι πεπισμένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει στην προσπάθεια αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λυθούν αυτά τα πράγματα και να συζητηθούν και γρήγορα και επικοδομητικά. Θα χρειαστεί όμω χρόνο και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε χρόνο. Εμεί πρέπει να δράσουμε τώρα. Πριν από μια εβδομάδα ήμουν στην Ιδωμένη και δεν ξεχνάω αυτέ τι εικόνε που είδα. Ήταν φρίκι αυτά που είδα. Ο κόσμο είναι απελπισμένο. Ε, ε, δεν έχουν στέγη, Κυρίω γυναικόπαιδα. Υποφέρουν εκεί. αυτέ τι εβδομάδε και τούτη εδώ τη η κατάσταση επιδεινώθηκε έτσι περαιτέρω. Με καταιγίδε, με νεροποντές. Με στη λάσπη είναι ο κόσμος και σήμερα ε, ε, μου είπαν ότι είναι 15.000 οι άνθρωποι στην Ιδωμένη, με πήραν τηλέφωνο και ζητούν ε, ε, βοήθεια. Η κατάσταση κινδυνεύει να εκραγεί. Κύριε Αβραμόπουλε, σα είπα από το Σεπτέμβριο την κατάσταση, σα έχω στείλει επιστολή, έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα σε σχέση με αυτό. Αν δεν υπήρχε ο ντόπιο πληθυσμό, η κατάσταση θα είχε εκραγεί εδώ και καιρό. Τώρα επιτέλου έχουμε ένα κανονισμό του Συμβουλίου, ένα νομικό πλαίσιο και σα εκλυπαρώ, πέφτω στα πόδια σα να δράσετε. Δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Χρειάζεται δράση διαπλασιάσει οπωσδήποτε. Όπως ε, έκανε και η πορτογαλική κυβέρνηση που θέλει να διαπλασιάσει την ποσόστοσή τη. Και από χτες οι πρόσφυγες φεύγουν από την Ελλάδα και πάνε στην Πορτογαλία. Αυτή είναι η σωστή απάντηση σε αυτή τη δύσκολη κρίση που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε μπλε κάρτα από τον κύριο Άτκινσον. Όχι, ήταν μπλε κάρτα, λέει η κυρία Άτκινσον για τον κύριο Μπροκ. Κύριε Μπροκ, δεν ε, θελήσατε να απαντήσετε στην ερώτησή μου. Την Κυριακή, όταν η κυρία Μέλκερ προσπαθούσε να καθησυχάσει ε, τον κύριο Ερντοάν, τι είπε για τα όσα έγιναν με τη Ζαμάν. Μίλησε για τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα των δημοσιογράφων οι οποίοι έπεσαν θύμα επίθεσης προχτές. Με τον κύριο Νταβούτογλου το είπε αυτό και με τον κύριο Ερντογάν τα έχει συζητήσει νη φορές. Ε, δέχεται πάντα επιθέσεις η κυρία Μέρκελ επειδή είναι πολύ σκληρή με την Τουρκία. Τα θέτει υπόψη την ελευθερία της ε, έκφρασης της θρησκείας και τα λοιπά. Σε αυτό το θέμα είναι πρωταθλήτρια η κυρία Μέρκελ ε, στην Τουρκία. Και για τα κεφάλαια 22-23 νομίζω είπε ότι θα πρέπει να, να ανοίξουν για να μιλάμε για την ελευθερία του τύπου, της θρησκείας και της έκφρασης που είναι προϋπόθεση για να ε, μπει η Τουρκία που απέχει πόρο και απέχει πολύ περισσότερο από ποτέ ε, με βάση τα τελευταία γεγονότα και σας διαβεβαιώ ότι αυτή είναι και η θέση της κυρίας Μέρκελ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, έχουμε κανόνες εδώ και θα πρέπει να τους σεβόμαστε στη διαδικασία. Όταν ζητείτε το λόγο για μπλε κάρτα, μετά από δύο μιλητές, δύο μιλητές αργότερα, παραβιάζετε τους κανόνες. Υπάρχει κανονισμό. Δεν σας είδε κανείς κύριε Άτκινσον να ζητείτε το λόγο την ώρα που μιλούσε ο κύριος Μπροκ. Και παρακαλώ να μην διαμαρτύρεστε. Και δύο μιλητές μετά κάνετε ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη κύριε Βάιντενφέλτσερ. Ε, και κυρία Άτκινσον την άλλη φορά δεν θα σα δώσω το λόγο. Κύριο Χαλάχο. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη στην αντιμετώπιση της, ε, του μεταναστευτικού. Ο μηχανισμός επανεγκατάστασης που έχει αποτύχει αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα κάποιο θέματος που προσπαθεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν ενδιαφέρει ούτε τις κυβερνήσεις ή τους μετανάστες. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι να κάνουμε το asylum shopping, δηλαδή να έρχονται οι άνθρωποι στην Ελλάδα και μετά χωρίς κανένα εμπόδιο να μπορούν να φεύγουν για τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Τώρα έχουν μειωθεί λίγο οι ροές, όχι γιατί έκανε κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τα κράτη-μέλη έχουν ξαναστήσει τους ελέγχους στα εσωτερικά ε, σύνορα. Θα πρέπει να ανασταλεί η Σέγγεν μέχρι η κατάσταση να ελεγχθεί. Διαφορετικά θα χαθεί η Σέγγεν τμήμα-τμήμα και θα πρέπει οι κανόνες για το άσυλο να ε, ξαναδιατυπωθούν έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να υποβάλει έτσι ασύλου για ένα κράτος αν έχει καταφτάσει σε άλλο. Ευχαριστώ κυρία Ναταλή Γκρίσπεκ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε σαν το μύθο του Σιζήφου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάλαβε επιτέλους για ποια κρίση πρόκειται και μετά από τρεις δέσμες δράσεις, αναθεωρήσεις, αξιολογήσεις και συνόδους κορυφής σήμερα ε, ε, πραγματικά είναι ε, κάτι που χωλαίνει η εφαρμογή για να μην πω ότι είναι απελπιστική. Γιατί εσείς κάτι χτίζετε το πρωί και το βράδυ τον κρεμίζουν οι κυβερνήσεις. Χρόνια ολόκληρα ζητούμε από το Κοινοβούλιο προστασία των εξωτερικών συνάρων για να προστατευτεί το Σέγγεν. νόμοι μεσοδούς και διάβλους για αλληλεγγύη στις χώρες. Όσο περνάει ο χρόνος τόσο λιγότερο αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι χώρες με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ελλάδα οι χώρες ε, πέφτουν σε μια διπλή παράλυσία ε, θανατηφόρα σε δύο επίπεδα. Πρώτον, γιατί ε, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα και εκατομμύρια οικογένειες καταστρέφονται από πολέμους και κατά δεύτερο λόγο τι παρατηρούμε και μάλιστα με σταυρωμένα τα χέρια στο ναυάγιο των αρχών που έκτισαν την Ευρώπη αντί για σύσυφη γίνεται προμηθής παρακαλώ κύριοι και φέρετε τα κράτη-μέλη ενώπιον των ευθυνών τους. Ο κύριος Χρυσόγονος παρακαλώ. Έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Έδειξε για μια ακόμη φορά ότι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένα κράτη-μέλη που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις κοινέ ευθύνε και δεν επιδεικνύουν αλληλεγγύη απέναντι στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ένα μείζον πανευρωπαϊκό πρόβλημα όπως είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό. πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μονομερείς ενέργειες και οι εγωιστικές εθνικές πολιτικές όχι μόνο δεν αποδίδουν αλλά μακροπρόθεσμα θα έχουν καταστροφικά αποτελέσματα για όλους. σημειώνω πάντως με ικανοποίηση τη δέσμευση της συνόδου για επαναπροώθηση στην τουρκία όσων εισέρχονται αυθαίρετα στο ελληνικό έδαφος και για κατανομή ίσου αριθμού σύριων προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη. επίσης καλωσορίζω την υπόσχεση για άμεση οικονομική και οργανωτική βοήθεια προς την ελλάδα ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των εγκλωβισμένων προσφύγων καθώς και για υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασής τους από την ελλάδα στα άλλα κράτη μέλη. τα λόγια όμως πρέπει να γίνουν έργα άμεσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαλέρο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ανησυχώ. Ανησυχώ πάρα πολύ για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το μέλλον της Σέγγεν. Φοβάμαι πως όλα αυτά θα καταρρεύσουν. Χώρα-χώρα. Κάθε χώρα αυτή τη στιγμή ξαναστείνει ελέγχου στα σύνορα προσωρινά και αυτό σε εισαγωγικά και αυτό συμβαίνει και με τη χώρα μου. Νομίζω πως δική μας δουλειά είναι να είμαστε ε, συνετοί και να ε, επαγρυπνούμε έτσι ώστε αυτοί οι ελεγχοί να διαρκέσουν όσο το δυνατόν λιγότερο. Όσο τα κράτη-μέλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, πάντα θα υπάρχουν έλεγχοι στα σύνορα. Και αυτό είναι τραγικό. Επίσης, συζητάμε για την επιστροφή όσων δεν χρήζουν άσυλο. Δεν είμαι επί της αρχής αρνητική, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που βρίσκονται στην Ευρώπη εδώ και χρόνια και έχουν ήδη λάβει ε, δια, ε, διαταγές επιστροφής και δεν έχουν επιστρέψει γιατί οι χώρες τους είναι πολύ επικίνδυνες. Έχουμε τη Λωρίδα της Γάζας, έχουμε το Αφγανιστάν. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Κύριος Μαρούση, κανένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι μας. Όλοι μας κάποιες φορές αρρωσταίνουμε. Άλλοι είμαστε γιατροί. Τι λέμε κάθε φορά. Πως είναι η ρίζα της ασθένειας θα πρέπει να καταπολεμηθεί και όχι τα συμπτώματα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι το αντίστροφο. Αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα και όχι την ίδια την ασθένεια. Νομίζω πω αν συνεχίσουμε έτσι θα καταστρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν νοιάζεται κανεί για τη Σέγγεν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει καταρχήν να ορίσουμε τι είναι η Ευρώπη και τι δεν είναι η Ευρώπη. Να κλείσουμε τα σύνορά μα και να αρχίσουμε να πολεμάμε κατά της εισρωής αυτής της ε, μόλυνσης. Δεν θα πρέπει να ε, κοιτάξουμε την ασθένεια και να τη στηρίξουμε και να τη βοηθήσουμε γιατί θα μας καταστρέψει. Η Τουρκία θα μας χρησιμοποιήσει. Θα πάρουν δισεκατομμύρια ευρώ για να εφαρμόσουν τις δικές τους πολιτικές και εμεί είμαστε ανίκανοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μα και να κλείσουμε τα εξωτερικά μα ε, σύνορα. Να αντιδράσουμε πιο ριζοσπαστικά προτείνω. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκάμπριελ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση όσον αφορά αυτό το θεματολόγιο. Όσον αφορά επίση την κινητοποίησή σα ε, από τότε που άρχισε η εντολή σα εμεί, το γνωρίζουμε ότι έχετε ακόμα πολλά να κάνετε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κύριε Επίτροπε. Τώρα έχω τι εξή ερωτήσει. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά την ε, συγκρότηση των hot spot, γιατί έχουμε πάρα πολλά τα οποία ακόμα δεν είναι λειτουργικά. Ποια είναι η βασική φραγμή, τα βασικά εμπόδια που μα εμποδίζουν να προχωρήσουμε ε, ταχύτερα. Αν είναι πολιτικό το θέμα, τότε θα πρέπει να κάνουμε περισσότερε προσπάθειε, ώστε να ληφθούν οι αποφάσει σε εθνικό επίπεδο. Και έτσι θα πρέπει ε, να μην αναβάλουμε για, για αύριο αυτό το οποίο είναι σημαντικό σήμερα. Γιατί αυτό το οποίο σήμερα αναβάλουμε θα γίνει αύριο κάτι κατεπίδευτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σα είπαμε ότι στον Ήγηρα έχει ε, αυτό το, το πιλωτικό σχέδιο. Ακόμα δεν έχουμε μάθει με αυτό το κέντρο πιλότο στον Ήγηρα. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε πώ θα διαμορφωθεί η εξωτερική πολιτική μα για το μεταναστευτικό. Θα πρέπει αυτό το project να το χρησιμοποιήσουμε τόσο ώστε να συνεργαστούμε με τι τρίτε χώρε, ιδίω τη Αφρική. Οπότε ε, κάτι άλλο για, το, ε, για την πολιτική μα το μεταναστευτικό θα πρέπει, σας τονίζω, να δούμε ότι θα πρέπει να φροντίσουμε το τι γίνεται εκτός συνόρων και έτσι θα αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες στο εσωτερικό. Ε, τι γίνεται με την επανεισδοχή. Ε, τι γίνεται με την ε, Ιορδανία. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και το Λίβανο και την Ιορδανία που είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται αυτό. Γιατί έχουμε ε, τι υποχρεώσει ή τι υποσχέσει οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πράξει. Κύριε Ροντρίγκης, έχετε το λόγο. Ναι, και εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ ε, τις τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά η ελληνική λύση και η τουρκική λύση ε, θα αποδειχθούν ότι έχουν τα όρια τους. Επομένως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ευρωπαϊκές λύσεις ώστε να πανακτήσουν την έλεγχο κατάσταση και θα πρέπει να προστατεύσουμε το Σέγγεν. Θα πρέπει επίσης να κάνουμε κάτι για τους ε, πρόσφυγες, χρειάζεται σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό σύνορο, όχι ε, σειρματοπλέγματα. Αυτό που χρειάζεται μια νέα σύλληψη ε, συστήματος συνόρων. Ε, θα πρέπει να έχουμε ε, υποδομές νέας γενιάς, να υπάρχει απαραίτητη υποδομή και επιμελητία, να υπάρχουν οι αντίστοιχε υπηρεσίες, ο έλεγχος, η διαχείριση των ροών και επίσης θα πρέπει να βοηθούμε με ευρωπαϊκά στάνταρ τους ε, πρόσφυγες, να οργανώσουμε, να χρηματοδοτήσουμε, να προωθήσουμε τέτοιες ε, ε, λύσεις, στρατηγικές επενδύσεις του δημοσίου. Αυτά θα πρέπει να στήσουμε, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι για τον 21ο αιώνα η Ευρώπη και έτσι να δούμε με πιο θετική άποψη τις εξωτερικές μας σχέσεις. Η Πρόεδρος, ο επόμενος αγορητής είναι η κύριε Φωστόρχη, Ευχαριστώ πολύ κύριε και Θα ήθελα να εστιάσω σε ένα κεντρικό ζήτημα του θεματολογίου για τη μετανάστευση, το μηχανισμό ανακατανομής. Εκατομμύρια είναι αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη. Ο Υπουργός Μούλερ ε, ανάπτυξη της Γερμανίας μίλησε για 8 με 10 εκατομμύρια από τη Μέση Ανατολή που είναι καθοδόν ήδη και από την Αφρική ακόμα πολύ περισσότερα εκατομμύρια θα μας έρθουν. Και ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει εδώ και μήνες για την κατανομή 160.000 από την Ελλάδα και την Ιταλία. 800 τόσοι ήδη έχουν μετακομίσει και τώρα μας λένε ότι θέλει επιτάχυνση. Άρα μήπως μόνο 15 χρόνια θα χρειαστούν για τις 160.000 που είναι εδώ παρόντες. Μα αυτοί πόσοι είναι, ε, θα έχουμε άλλα 10 ή 20 εκατομμύρια που θα σειρεύσουν. Τι σχέση έχουν τα μεγέθη αυτά μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε όλους στην Ευρώπη. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε στον τόπο τους και μάλιστα αμέσως, τώρα. Ευχαριστώ κυρία Αλμπιόλ. Γκουσμάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Οι μεταναστευτικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίχθηκαν ανάλογα με τις επιταγές της οικονομίας ή τουλάχιστον της οικονομίας κάποιων και πάντα στο περιθώριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ξεκίνησαν μοιράζοντα τους μετανάστες σε δύο ομάδες, παράνομοι και νόμιμοι. Στους παρανόμους έχτισαν τύχη, τους έκλεισαν σε κέντρα, τους αφαίρεσαν την πρόσβαση ε, στα νοσοκομεία, ε, κάνανε αποθήσεις εν θερμό και μετά από τους πολέμους στο Αφγανιστάν, στη Συρία και στο Ιράκ χρησιμοποίησαν με φρικτό τρόπο τους πρόσφυγες για να ξεχωρίσουν τους πρόσφυγες από τους μετανάστες. Είπανε είναι οικονομικοί μετανάστες. Άρα λοιπόν οι πρόσφυγες έχουν κάποια δίκιο μετά οι μετανάστες. Κανένα. Όλοι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ούτε αυτό. Τώρα και οι πρόσφυγες θα διώχνονται στα σύνορα ή θα τους αφήνουν στα στρατόπεδα του καλέ χωρίς καμία αξιοπρέπεια. Όλοι, όλες οι πρόσφυγες, οι μετανάστες είναι τα θύματα των ε, σκληρών σας και κοινικών σας πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μαραγκάλ. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται πως το σημείο αφετηρίας είναι να περιορίσουμε, να αποφύγουμε και μετά να αρνηθούμε, να επιστρέψουμε και να επαναπατρίσουμε. Και μετά συμφωνίες με τον σατανά τον ίδιο, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε απευθείας τα προβλήματα. Το κάναμε αυτό. Αυτή είναι η, Ευρωπαϊκή, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έχουμε το πλαίσιο που περιγράφει η σύμβαση του Δουβλίνου αλλά αυτή η μεμονωμένη αντιμετώπιση των ετοιμάτων ασύλου έμεινε πια στην ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Ελλάδα που είναι στο χείλος της Αβίσου και που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ή τεράστιο ε, σοφρονιστικό κέντρο ή ως δοχείο στο οποίο θα παρκάρουμε ανθρώπους. Κλείνουμε ε, την οδό των Βαλκανίων και δεν μπορούμε εμείς τα κράτη-μέλη να αλλάξουμε κάτι. Και παιδιά, γυναίκες, άντρες... Ε, ίσα ίσα επιβιώνουν συνειδωμένοι. Υπάρχουν κάποια εθνικά συμφέροντα τα οποία προωθούμε και έχουμε ξεχάσει τα ευρωπαϊκά. Η απόκριση που πρέπει να δώσουμε να αλλάξουμε τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε, όχι αυτό που προτείνεται. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχετε χρόνο, όσο γρήγορα και να μιλήσετε, δεν θα σας ακούσει κανείς. Η κυρία Άτκινσον. Ε, ξέρετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα καταφέρνει καλά στα παζάρια όταν πάει στα παζάρια τα τουρκικά. 20 δι ζήτησε η Τουρκία. Μα με συγχωρείτε, πόσο πια θα δώσετε από τα χρήματα του φορολογωμένου. Και μετά ο κύριο Στάρκ στο στο αεροπλανό, αφού ε, συμφώνησε για τον οδικό χάρτη, ε, είδε ότι κλείσαν τη ζαμάν. Και η κυρία Μέρκελ μα είπε την Κυριακή η... πως το πιο σημαντικό είναι ε, τι θα πούνε οι εκλογείς. Έχετε ακούσει τη γνώμη των ε, Ευρωπαίων. Θέλουν να απελευθερώσουν τις θεωρήσεις για 75 εκατομμύρια Τούρκους. Έχετε ακούσει τους Βρετανούς αν θέλουν να πληρώσουν άλλα 150 δις στα 12, δις, στα 12 που πληρώνουμε ήδη. Δεν νομίζω. Αν λοιπόν μου πείτε τι κερδίσατε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις στο τουρκικό παζάρι, νομίζω πως δεν κερδίσατε πολλά, σας κορόιδεψαν και οι Βρετανοί αυτό θα το διορθώσουν. Ευχαριστώ, Δίας Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τονίζω τη σημασία των αριθμών, των αφήξεων. Αντιμετωπίζουμε ανθρωπιστική κρίση τεράστια και κρίση διαχειριστική επίσης. Θα πρέπει να τερματιστεί η μονομερής ε, ε ενέργεια ε, του κλεισίματος των συνόρων. Όπως και ο Φίλιππο Γκράντι θέλω και εγώ ανοιχτά τα Βαλκάνια. Μόνο με αλληλεγγύη θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη σκληρή κατάσταση. Θα πρέπει να επανέλθει η Σέγγεν και να την προστατεύσουμε με περισσότερο έλεγχο στα εξωτερικά όμως σύνορα. Στηρίζω τα επίγοντα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το μηχανισμό ανθρωπιστικής βοήθειας επίσης επίγοντα για την Ελλάδα και την επίγουσα αποστολή των ε, όσων ε, από τα ποσά από τα άλλα δύο ταμεία για την Τουρκία. Αυτό είναι ένα θέμα δύσκολο. Η Τουρκία τώρα, ναι, αλλά γιατί. Για να βελτιωθούν οι ανθρωπιστικές συνθήκες ε, στην επικράτεια της Τουρκίας για τους πρόσφυγες και στη Συρία. Και η Τουρκία χρειάζεται για να φρενάρει τις ροές εκείνων που δεν χρειάζονται διεθνή προστασία. Δεν έχουμε και υπερβολικά πολλές εναλλακτικέ. Θα πρέπει να αντιποκριθούμε στις εσωτερικές και εξωτερικές υποχρεώσεις. Επανεγκατάσταση, μετεκατάσταση, hot spots και ε, πόρους. Και ο ακρογωνίος λήθος διεθνώς ποιος είναι να τηρηθεί το ψήφισμα 2268 για την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Να επανειληφθούν και να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες της Γενέβης. Τελειώνω, Πρόεδρε. Και οι δύο ομάδες εργασίες, κυρίως ε, που είμαστε εκεί πάρα πολύ σημαντικοί και πάρα πολύ αξιόπιστοι. Αυτά τα ολίγα και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Γιώτοβα. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω να σας στηρίζω ναι, έτσι να αντιμετωπίσετε την κρίση. Όμως θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν έμπαινε πολύ αισιοδοξία η προηγούμενη ζήτηση για την Συρία. Έχουμε δύο άξονες εδώ, δύο πυλώνες. Πρώτα-πρώτα την επίλυση, για αντιμετώπιση των ε, συγκρούσεων αλλά και τη διαχείριση των κρίσεων. Ε, τώρα τελευταία ασχολούμαστε μόνο με το δεύτερο. Δεν έχουμε συνολική σφαιρική πολιτική για τη μετανάστευση σήμερα. Ε, είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε στενά περιφερειακά το, το θέμα της ε, διαχείρισης των νερών. Τώρα ε, αναδύθηκε το θέμα της Ελλάδος, το θεματολόγιο. Η κατάσταση είναι έκτακτη. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί όλες σας οι προτάσεις κατατείνουν στο να περισωθεί το Σέγγεν. Το Σέγγεν είναι τώρα τη μόδα όμω. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα σύνορα. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα σύνορα. Ε, ουδέτερη ζώνη, νεκρή ζώνη, θα γίνουν και, και εκεί ένα μεγάλο στρατόπεδο. Δεν θα έχουμε καμία ασφάλεια μετά. Η πρόοδο. Για ένα λεπτό, κύριος Ουγιασντόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι θα πρέπει να περτανεύσει και πάλι ο ρεαλισμός. Όχι ο λακισμός, ο ρεαλισμός, διότι πέρυσι όλοι ανέφεραν για την πολιτική των ανοιχτών συνόρων. Αυτό ήταν μάλλον ανεύθυνο. Άρα χαιρετίζω την επάνωδο στον ρεαλισμό, να υπάρξει έλεγχος των συνόρων, να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Αλλά θα πρέπει να απαιτηθεί να είναι αξιόπιστη, να είναι υπεύθυνη η Ελλάδα τελική συμφωνία με την Τουρκία να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες, τους χριστιανούς, αλλά και τους υπολείπους αυτοί οι οποίοι υποφέρουν από τον πόλεμο. Να ξαναγυρίσουμε ε, στο θέμα της ε, μετεγκατάστασης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό το σύστημα είναι κάπως επικίνδυνο ε, δεν είναι δυνατόν να μετακομίζουμε τον κόσμο κάπου που δεν θέλουν να πάνε. Ας βοηθήσουμε τον κόσμο. Κύριε Σακοράφα, τώρα έχει το λόγο. Όποιο θέλει να κατανοήσει την κατρακύλα τη Ενωμένης ΕΕ Ευρώπης και των ηγετών τη, αρκεί να διαβάσει τα συμπεράσματα τη χθεσινή Συνόδου Κορυφή. Η Ενωμένη Ευρώπη των αρχών και των αξιών στη σκληρή διαπραγμάτευσή τη με την Τουρκία, το κράτο που παραβιάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, κατέχει με στρατό ευρωπαϊκό έδαφος παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες βομβαρδίζει εντός και εκτός συνόρων τις κούρδους πολίτες και ο πρόεδρός της εκβιάζει με την απελπισία χιλιάδων προσφύγων πέτυχε την απαλλαγή της βίζας το άνοιγμα ενταξιακών κεφαλαίων την εκταμείευση τριών δισεκατομμυρίων και επιπρόσθετης χρηματοδότησης και το κορυφαίο που είναι ντροπή ακόμα και να γράφεται την ανταλλαγή έναν προς έναν πρόσφυγα παράλληλα έχει ήδη πετύχει να κλείνουν σύνορα κατά το δοκούν να μετατραπεί η ελλάδα σε καταβλισμό δυστυχισμένων και να εξαργυρώσει το αμόλυντο της ησυχίας της με κατακεφαλήν ποσά για κάθε πρόσφυγα καταργώντας στην πράξη το άσυλο και παραβιάζοντας διεθνείς συνθήκες. και επέρονται ομού γερμανική αυστριακή και ελληνική ηγεσία. δυστυχώς κύριοι συνάδελφοι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και τραγικές. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ρεμπέγκα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει εξαγγείλει κάποιες δράσεις. Τώρα ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αρχή της αλληλεγγύης ε, και οι συγκεκριμένες προτάσεις. Τι να τα κάνουμε όλα αυτά τα σχέδια δράσης ε, όταν δεν εφαρμόζονται. Κινδυνεύει η Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μια μεταναστευτική πολιτική με σταθερότητα και με βάση τη σύμβαση του Δουβλίνου. Αυτή είναι απόλυτη προτεραιότητα κανονικά. Οι ε, ηγέτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δείξουν ηγετική στάση. Χρειάζεται οπωσδήποτε δράση και όχι αυτά τα ουτοπικά που ακούμε. Είναι πολύ ε, λίγα αυτά που ε, κάνουμε. Έχουμε πέσει σε λίθαργο, μας λείπει κοινή εικόνα, κοινό όραμα και είναι εις βάρος όλης της Ευρώπης αυτό. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Σβέρ. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Συνάδελφοι, στηρίζω τα συμπεράσματα της εκτάκτου Συνόδου Κορυφής. Δυστυχώς η Ευρώπη χτες το βράδυ βγήκε για ψώνια. Αγοράσαμε υποσχέσεις πως οι ροές μεταναστών θα ανασταλούν ή τουλάχιστον θα επιβραδυνθούν και τελικά πως θα ξαναστηθεί η Σέγγεν. Και αγοράσαμε σε πολύ ακριβές τιμές, ειδικά αν η Τουρκία σταθεί αναξιόπιστος εταίρος. Οι αποφάσεις οι οποίες θα παρθούν την επόμενη εβδομάδα ελπίζω να είναι πιο λογικές και τότε ενδεχομένως η κατάσταση θα βελτιωθεί. Δεν έχουμε εξασφαλίσει μόνο πολύ επιπλέον οικονομική στήριξη για την Τουρκία. Δώσαμε και υποσχέσεις για μια διαδικασία ένταξη επιταχυμένη. Παρόλο που αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με τη μεταναστευτική κρίση. Αισθάνθηκε την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τουρκία και μας εκβίασε. Δεν είναι αξιόπιστος εταίρος. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή που αποδεικνύει θετικό πνεύμα. Και αυτό βεβαίως δημιουργεί ανησυχίες για το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκία. Σήμερα με ρώτησε κάποιος δημοσιογράφος και τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί έχουμε δημοσιογράφους στην Τουρκία για τους οποίους ανησυχούμε. Και μετά από τη χθεσινή σύνοδο Κορυφή, ελπίζω πω κάτι θα έχετε ξεπεράσει το χρόνο σα συνάδελφοι. Η κυρία Σλάιντ είναι η επόμενη ομιλήτρια. Διακυβεύεται το μέλλον τη Ευρώπη, διακυβεύεται από το πώ θα μπορούμε να ε, ανταποκριθούμε. Έτσι θα μα κρίνουν οι επόμενε γενιέ. Παρ' όλα αυτά όμω συνεχίζουμε και μιλάμε, κάνουμε συναντήσει κορυφή και δεν φτάνουμε σε κάποια κοινή ευρωπαϊκή λύση το 2015 και πάντα είχαμε 6 από τους 28 ε, οι οποίοι είχαν το 80% των αιτήσεων ε, ασύλου. Αν είχατε κάνει αυτό που έπρεπε θα ήταν διαχειρίσιμη αυτά τα νούμερα ε, όπως και η Ιταλία και οι άλλες χώρες θα είχαν καλυφθεί αυτοί που κάνουν τις μεγάλες προσπάθειες. Το να κλείνουν τα σύνορα δεν είναι λύση οι κυβερνήσεις δεν θα είχαν υποστεί τον εκβιασμό της Τουρκίας. Κοινέ λύσεις με βάση την αλληλεγγύη και την σφαιρική προσέγγιση. Και σήμερα καθόμαστε και μιλάμε για την υλοποίηση του θεματολογίου. Μα πώς είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες μετακαταστήσεις που να γίνονται μόνο για κάποιες ε, ε, εκατοντάδες, αν έχουμε 150.000 μετανάστες. Είδατε τι έγινε στη Λαμπετούζα, εκεί που είχαν μπλοκαριστεί πάνω στο νησί ολόκληρες εβδομάδες ε, ούτε παπούτσια δεν είχαν και έχει αποδειχθεί επομένω ότι δεν μπορούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υλοποιήσουν τι αποφάσεις ε, του Συμβουλίου το οποίο οι ίδιες χώρες συναπαρτίζουν άρα χρειάζεται να υπάρξει μια προοπτική, ένα μέλλον το σύστημα των hot spot δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί φοβούνται αυτοί οι άνθρωποι να δεν ωφελούνται το Δουβλίνο είναι υποκριτικό χρειάζεται να αναθεωρηθεί με τολμηρά το Δουβλίνο και η Άσο επίσης να μεταρρυθμιστεί οπότε πάνω σε αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να μην είναι πια ο ρόλος μας ε, διακοσμητικός. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε αλλά δεν είναι δυνατόν να σας παρακολουθήσουμε αυτή την ταχύτητα οι διερμηνείς. Μιλήσατε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν περνάει το μήνυμα κύριο είναι ο που το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέτυχε να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση και συνεχίζει να λαμβάνει λαθασμένε αποφάσει που παραβιάζουν το ευρωπαϊκό και διεθνέ δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων. Πόσοι ακόμη πρόσφυγε πρέπει να πεθάνουν αβοήθητοι για να πάψουν οι ξενοφοβικέ ρατσιστικέ προσεγγίσεις ορισμένων Ευρωπαίων ηγητών όπως το χωρών του βισεγκράτ οι οποίοι κλείνουν τα σύνορα χτίζουν φράχτες και εγκλωβίζουν έτσι τους πρόσφυγες σε απάνθρωπες συνθήκες στην ελλάδα. κατάντησε το συμβούλιο να συζητά τις απαράδεκτες αξιώσεις και τους εκβιασμούς της τουρκίας για να αποφύγουν τα κράτη μέλη τις ευθύνες τους. και ας έχει η ευρωπαϊκή ε, ένωση ευθύνη για τους πολέμους που κατάστρεψαν τις χώρες των προσφύγων. το κλείσιμο του βαλκανικού διαδρόμου το νατο στο αιγαίο που καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών και τα κατασταλτικά μέτρα της frontex σκοτώνουν την αλληλεγγύη και τις αξίες της ένωσης. σταματήστε τη βαρβαρότητα. πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα νόμιμοι και ασφαλείς οδοί καθώς και ένα δεσμευτικό δίκαιο σύστημα κατάσταση των προσήγων. η προσφυγική κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενίσχυση της αλληλεγγύης που επιδεικνύει ο ελληνικός λαός. Ο κύριος Μπουονάνο, επόμενος μας. Είπατε να μιλάμε αργά, αλλά έχουμε ένα λεπτό. Μα πώ είναι δυνατόν να μπορέσουμε να, να, να, να κάνουμε έτσι μια ε, κουβέντα. Mm. Δεν έχω δίκιο. Τέλο πάντων. Ε, τι να κάνω τώρα, να το πω γρήγορα. Η Πρόεδρος. Μα, εγώ, λέει η πρόεδρος, προσπαθούσα να σας πω ότι ναι, όντως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορείτε αποτελεσματικά να μιλήσετε σε ένα ε, λεπτό. Οπότε μηδενίζω το χρονόμετρο, αρχίστε ξανά. Α, ωραία, μπράβο. Και σας ευχαριστώ, λέει ο κ. Μπονάνο. Άκουσα τα όσα κουβεντιάσαμε σήμερα και θέλω να σας πω ποια είναι η δική μου εμπειρία ως δημάρχου από κάποια τελική πόλη. Έφτασαν εκεί κάποιοι πρόσφυγες ε, και ούτε ένας από αυτούς δεν ήταν από τον πόλεμο. Ήταν από χώρες που δεν υπάρχει πόλεμος. Ε, θέλω να σας πω ότι τέλος υπάρχουν ε, πολλά και βέβαια είπαμε ότι άλλοι αποφασίζουν για την τύχη της Ευρώπης όπου κάθε χώρα ε, ε, έδωσε μάχη για να αποκτήσει την εξαρτησία της. Έχουμε τώρα όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι φεύγουν από τον πόλεμο και έρχονται στην ε, Ευρώπη. Είπαμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό είναι σωστό. Αλλά γιατί να μην τους ξαναστείλουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, στο, στην πατρίδα τους και εκεί να δώσουν τη μάχη για την εξαρτησία της χώρας τους. Λοιπόν, να τους δώσουμε ένα χεράκι για να διορθώσουν τα πράγματα στη χώρα τους. Να τους στείλουμε εκεί πέρα και εκεί να πολεμήσουν για την ελευθερία, την ανεξαρτησία της πατρίδας τους. Η Πρόεδρος, ο επόμενος ομιλητής, είναι η κυρία Βόζεμπεργκ στη χθεσινή σύνοδο κορυφής επί δεκαπέντε ώρες αναζητήθηκε το αυτονόητο ενώ οι οριστικές αποφάσεις αναβλήθηκαν για τις δεκαοκτώ του μηνός. αν όμως επί δέκα μέρες που απομένουν δυόμισι χιλιάδε περίπου πρόσφυγες και μετανάστες συνεχίσουν να έρχονται καθημερινά στα ελληνικά νησιά πώς θα αντιμετωπιστεί το ήδη τεράστιο αυτό ευρωπαϊκό τονίζω πρόβλημα με πρόσθετους είκοσι πέντε τριάντα χιλιάδες ανθρώπους; η ευρωπαϊκή ένωση έχει υποχρέωση και καθήκον να λάβει σοβαρέ αποφάσει για τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τι αποφάσει τη για μετεγκατάσταση προσφύγων στα εδάφη του να υλοποιήσει σε συνεργασία με την τουρκία επανεγκατάσταση προσφύγων από τα τουρκικά εδάφη απευθεία αναλογικά στι χώρε τη ευρωπαϊκή ένωση να σκληρύνει τη στάση τη απέναντι στι χώρε που αυθαίρετα κλείνουν τα σύνορά του και να υποχρεώσει την τουρκία να δεχθεί του παράτυπου μετανάστε που φιλοξενούνται στην ελλάδα τηρώντα επιτέλου επιτέλους υπογραφές της παλιότερες και πρόσφατες περί επανεισδοχής. αν συνάδελφοι ματαιωθεί οριστικά στην πράξη η οφειλόμενη αλληλεγγύη των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και αν η τουρκία ως στρατηγικός εταίρος εξακολουθήσει να προκαλεί συνεχώς με νέες απαιτήσει εκμεταλλευόμενη χιλιάδες απελπισμένους ανθρώπους η ευρώπη των αξιών και του ανθρωπισμού θα έχει οριστικά αποτύχει. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κυρία Πρόεδρε. Όσο εμείς συζητούμε εδώ και όχι για πρώτη φορά αυτό το θέμα, ταυτόχρονα στα σύνορα με τη Μακεδονία, λέει ο μιλητής, ε, παίζουν μέσα στις λάσπες προσφυγόπουλα και στους υπονόμους. Ε, έχουν πέσει όμοιροι οι πολιτικοί μας ε, στα χέρια λαϊκιστών και ακροδεξιών και νομίζουν ότι φράχτες με ηλεκτροφόρα σύρματα μπορούν και αγαθωτά σύρματοπλέγματα να λύσουν το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να γυρίσει πίσω και δεν μπορεί να συνεχίσει και το δρόμο του. Σκεφτείτε τις μητέρες που πήραν τη πιο δύσκολη απόφαση της ζωής τους όταν αποφάσισαν να φύγουν από τα σπίτια τους και να ζητήσουν μια καλύτερη ζωή. Τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μαζί με τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα βρουν μια καλύτερη ελπίδα και μια νέα πατρίδα για να μπορέσουν να αναθρέψουν τα παιδιά τους σε ειρήνη. Τα κλειστά σύνορα στην Ευρώπη είναι έσχος. Διαρριγνύουμε τα μάτια μας για τις αξίες μας και τον ανθρωπισμό. Η Ευρώπη δεν χρειάζεται προστασία από τους μετανάστες, αλλά από τους ίδιους τους μικρόψυχους πολιτικούς της που κοιτάνε μόνο τη σταδιοδρομία, την καριέρα τους και τα μικροπολιτικά και κομματικά τους ωφέλη. Δεν μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ε, χώρα μέλος που αρνείται να ε, εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, με αυτά που μας είπατε και με τα χτεσινά συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής αποδεικνύεται ότι η προσφυγική πολιτική της ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα παζάρι με την Τουρκία. Η Τουρκία αξιοποιεί την προσφυγική κρίση για να αναβαθμίσει το ρόλο της, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αμφισβητεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Από αυτά που αποφασίστηκαν χτες απομονώνω την συμφωνία ένα σου στέλνουμε ένα παίρνεις λες και ανταλλάσσουμε εμπορεύματα που είναι ό,τι πιο χυδαίο και ό,τι πιο διαστραμμένο έχει σκεφτεί ο ανθρώπινος νους. Κατά τα άλλα, κύριε Αντιπρόεδρε, παζαρεύεται αυτή την περίοδο με την Ελλάδα το χαλάρωμα της συζήτηση όσο αφορά τις δεσμεύσεις ή και την ελάφρυνση του χρέους προκειμένου η χώρα να μεταβληθεί σε ένα απέραντο hot spot καταστρέψατε τη χώρα με τρία μνημόνια και τώρα προσπαθείτε να την αποτελειώσετε με την προσφυγική κρίση. εντάξει θα υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια. αυτές οι συμφωνίες αποτελούν έγκλημα σε βάρος των προσφύγων ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι σήμερα στην ελλάδα και σε βάρος της χώρας. δυστυχώς αυτές οι συμφωνίες τις υπογράφει και η σημερινή κυβέρνηση τσίπρα. σας ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου. Πολλά μεγάλα λόγια ακούμε και λίγη δράση βλέπουμε το τελευταίο εξάμεινο. Η Ευρώπη αποσταθεροποιείται, η περιοχή ολόκληρη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Και αυτή η ε, ανεξέλεγκτη ε, ροή προσφύγων και μεταναστών θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τακτοποιήσουμε ε, αυτή την κατάσταση. Ακούμε για προσφυγική κρίση, αλλά ξέρουμε ότι μικρό κλάσμα αυτών των ανθρώπων είναι πρόσφυγες ή θα πάρουν το καθεστώς του πρόσφυγα. Είναι πολύ λίγοι εκείνοι που πραγματικά ζητούν άσυλο. Οι περισσότεροι δεν είναι καν πρόσφυγες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι απλώς παράνομοι οικονομικοί μετανάστες που αναζητούν μια καλύτερη ζωή, μια καλύτερη δουλειά, μια καλύτερη μοίρα. Γι' αυτό ε, υψοκινδυνεύουν και την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή των παιδιών τους δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τους δεχθούμε όλους αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματά της και ότι μπορεί να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα. Χρειάζεται και σαφείς δράσεις και δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Ευχαριστώ. Η κυρία Κιέγγε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, όσον αφορά το προσφυγικό, έχουμε μια σειρά προτάσεων που έχουν υποβληθεί. μερικέ από αυτέ τι ε, προτάσεις ήδη ε, προέρχονται από κοινοβούλιο, από ε, το Συμβούλιο. Τώρα επεξεργαζόμαστε και άλλε προτάσει, οπότε θα πρέπει να λάβουμε τι ευθύνε μα να προχωρήσουμε, αλλά χρειάζεται να τροποποιηθεί ο κανονισμό του Δουβλίνου. Γιατί ε, κατά αυτόν τον τρόπο δεσμεύει πάρα πολύ στην χώρα πρώτη υποδοχή των ετών άσυλο. Πρέπει να δοθεί μια ε, απάντηση. Η απάντηση μπορεί να έχει βάση μόνο την αλληλεγγύη, τον σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και επίσης τις αρχές του διεθνούς δικαίου τους γενικά αποδεκτές. Επομένως η ανθρωπιστική βοήθεια είναι μόνο ένα τμήμα μιας σφαιρικής προσέγγισης και στρατηγικής που εμείς στο Κοινοβουλίο το ζητούμε τόσο καιρό, τόσου μήνες χρειάζεται να βλέπουμε πιο μακριά ως Ευρώπη. αλλιώ. πάμε για ε, καταστροφή, για αποτυχία. Ε, σήμερα το πρωί τα συζητήσαμε και ε, είπαμε ότι θα πρέπει να σε στις αρχές πάνω σα οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοσλόφσκα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Κύριε Επιτροπή θα πρέπει να σας αναφέρω ε, κάτι το οποίο είπε, ζήτησε, πρότεινε ο κύριος Τούσκ για τους οικονομικούς μετανάστες. Τους είπε να μην έρχονται στην Ευρώπη. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ πρωτότυπο για την ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, τώρα που θα αντιμετωπίσει αυτά τα κύματα των μεταναστών, μιλάμε για πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος. Πώς να συνεχίσουμε έτσι. Πώς θα αναλάβουμε το άχθος αυτής της κρίσης θα πρέπει να έχουμε μια εξωτερική πολιτική, να σταθεροποιήσουμε Μέση Ανατολή και Αφρική. Και έτσι οι πρόσφυγες ή οι μετανάστες να μπορούν κάπου να επιστρέψουν. Άρα έτσι θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποια λύση. Είχαμε τη χθεσινή συμφωνία με την Τουρκία, είχαμε κάποιες λύσεις που χθε προτάθηκαν και έτσι υπάρχει κάποια ακτίδα ελπίδας ότι θα μπορέσουμε να μετακινήσουμε την προσοχή μας, ε, το κέντρο βάρους από την εσωτερική στην εξωτερική πολιτική πρέπει ομένω να αναλάβουμε το κόστος και όχι μόνο το οικονομικό γιατί βέβαια το τίμημα θα είναι πάρα πολύ υψηλό όσον αφορά το να αρχίσει η ελεύθερη διακίνηση προσώπων με την Τουρκία. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά είναι σημαντικά για την ασφάλεια αλλά θα είναι σημαντικά και για να μπορούμε αποτελεσματικά να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες θα πρέπει να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε επί τη βάση στοιχείων αξιόπιστων, να δούμε τι πρέπει να γίνει ακριβώς, να υπολογίσουμε τις διάφορες δαπάνες, να δούμε τι μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να μην πλημμυρίσουμε και να είναι πάρα υπερβολική επιβάρυνση αυτής της αρρωγής. Κύριε Κύρκο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό το κοινοβούλιο πάντα αναζητούσαμε τους νόμους και ασφαλείς τρόπους εισρωής των προσφύγων στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, στη χθεσινή ανακοίνωση, βλέπουμε ένα ψήγμα από αυτό το δρόμο, που είναι ο μηχανισμό τη επανεγκατάσταση από την Τουρκία κατευθείαν στην Ευρώπη. Αυτό συνδυαστεί μαζί με τη μετεγκατάσταση όσων προσφύγων είναι στην Ελλάδα σε ευρωπαϊκέ χώρε και με την απόλυτη επιστροφή όσων είναι οικονομικοί μετανάστε στην Τουρκία και από εκεί στι χώρε του, μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ε, να προσεγγίζουμε μια λύση του προβλήματο. Ποιο είναι όμω το κόστο που πληρώνουμε γι' αυτό το κόστος δυστυχώς είναι η έκπτωση που κάνουμε στις αξίες μας, η έκπτωση στις αρχές μας, κυρίως αυτές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι το αντίτιμο που πληρώνουμε γιατί δεν προχωράμε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, δεν προχωράμε στην πολιτική ενοποίηση δίπλα στην οικονομική. Αυτό είναι το κόστος που μας βάζει να πληρώσουμε η Επιτροπή, η οποία μας είπε ο κύριος Γιούνκερ πως είναι Επιτροπή τελευταίας ευκαιρίας. Ζητάμε από τους Επίτροπους να κάνουν το καθήκον τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Μογανό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα δεν ευθύνεται για την ε, μεταναστευτική τραγωδία που ζούμε στην Ευρώπη. Αλλά με την ασυνάρτητη πολιτική της και τα μηνύματα που έστειλε, ε, προκάλεσε κατά πολύ τη λαθρομετανάστευση στην επικράτειά της. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώνουμε ότι όταν ακούνε για ποσοστώσεις, οι μετανάστες ενθαρρύνονται να έρχονται στην Ευρώπη. Η πραγματικότητα ποια είναι. Στη Γαλλία η κυβέρνηση επέλεξε να ε, αδειάσει αυτή την απαράδεκτη και αναξιοπρεπή ζούγκλα στο Καλέ για να τους στείλει σε διάφορα χωριά στη Γαλλία. Και στο χώρο Σέγγελ, σε ε, αυτά τα κέντρα υποδοχής ε, δεν έχουμε σύνορα και δεν είναι και φυλακέ κλειστά κέντρα. Και πάνω από το 1 τέταρτο των μεταναστών που εστάλησαν σε αυτά τα χωριά έφυγαν χωρίς να ξέρουμε πού βρίσκονται. Και στην Γερμανία 160.000 άνθρωποι κυκλοφορούν γενικά χωρίς να ξέρουμε πού βρίσκονται. Ορισμένοι από αυτούς έφτασαν και στη Γαλλία και στη δική μα επικράτεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποκτήσουν στον ήλιο μοίρα. Και εμείς ε, τους προσελκύσαμε με ψεύδι. Αυτή είναι η συναρτησία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η σημερινή πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον. Χρειάζεται σθένος στην πολιτική. Να στείλουμε ένα μήνυμα και με πολιτική επιστροφών που δεν έχουμε σήμερα, διότι σήμερα η μεταναστευτική πολιτική είναι ε, απολύτως ε, έρμεο της κατάστασης. Πρέπει να το καταλάβουμε στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Σεσχόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πριν ξεκινήσει ο χειμώνα, οι περισσότεροι από εμά θεωρούσαμε πω τα κύματα των μεταναστών και των προσφύγων θα μειωθούν λόγω του καιρού και ίσω θα σταματήσουν κιόλα. Αυτό δεν συνέβη. Και τώρα η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγαλύτερο ε, πρόβλημα από ό,τι πέρσι τέτοια εποχή. Έφτασε η ώρα να καταλάβουμε πω έχουμε πιο πολλά προβλήματα από ό,τι φανταζόμασταν. Ήμουν σε θέση να δω με τα ίδια μου τα μάτια πως η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει τη ροή των, προσφύγων και κυρίως την κατάσταση με στα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Μακεδονίας, λέει ο μιλητής. Ώρα ήρθε αυτό να αλλάξει. Και αν δεν γίνει κάτι γρήγορα, η Ελλάδα δεν θα μπορεί πια να προστατεύσει την περιοχή Σέγγεν. Και αν αυτό συμβεί, δεν θα μας βοηθήσει τίποτα. Ας μιλήσουμε πρώτα για συγκεκριμένα μέτρα. Ας μιλήσουμε πρώτα για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε μεταξύ Βαλκανικών χωρών, εταιρική σχέση με την Τουρκία, δημιουργία μιας ε, ακτοφυλακής ε, και συνοριοφυλακής ευρωπαϊκής. Αυτά είναι τα εργαλεία τα οποία παρόλα αυτά δεν μπορούν από μόνα τους να μας σώσουν εφαρμόσουν. Κύριος ευχαριστώ Πρόεδρε. Για πολλωστή φορά βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε το θέμα της μετανάστευσης και συζητούμε όλα αυτά τα κατεπήγοντα που έχουν εμφανιστεί και εγώ σας λέω θα πρέπει άπαξ ε, και διαπαντός να σταματήσουμε τα λόγια και να αρχίσουμε τα έργα και το πιο σημαντικό σημείο είναι το πώς θα τροποποιηθεί η τρίτη συνθήκη του Δουβλίνου. Πρώτα για μια ανομαλία στο σύστημα υποδοχής και έτσι θα μπορέσουμε με συγκεκριμένο τρόπο να βοηθήσουμε σήμερα την Ελλάδα, αύριο την Μάλτα, χθε να έχουμε δει στην Ιταλία ή αύριο την, μεθαύριο την Ισπανία τέλο πάντων. Θα πρέπει, είπαμε, μέχρι τις 31 Τρίτου να έχει κατέβει πρόταση για την τροποποίηση της συνθήκης. Ε, θα πρέπει να τηρηθεί όμως αυτή η καταληκτική ημερομηνία και αυτό που θα σας πω είναι ότι ε, τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να φερθούν υπεύθυνα και με συνέπεια. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κύριε κορατσομπίλτ, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, τα κλειστά σύνορα και οι ποσοστώσεις μεταθέτουν σε άλλο κράτο μέλος το βάρος. Θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία, θα πρέπει ε, να έχουμε κάποια έφτακτη υποδοχή και ασφάλεια στα σύνορα και να φερθούμε ανθρώπινα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει επίσης το ΣΕΝΙΑ ξανασταθεί στα πόδια θα πρέπει να έχουμε μια βάση δεδομένων. Ε, έτσι να γίνει συνεργασία με την Τουρκία. Είμαι υπέρ αυτής της συνεργασία, να υπάρξει ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ελλάδα ε, να βοηθήσει η Τουρκία, η Ιορδανία αλλά και Λίβανο και να εκταμιευθούν ταχαίω οι σχετικοί πόροι να βοηθήσουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και ο ΙΕ ε, είμαι υπέρ του ΝΑΤΟ να βοηθήσει ε, στο Επίση θα πρέπει από όλα τα κράτη-μέλη να υπάρχει ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων, να ξαναδούμε τις ποσοστώσεις, να δούμε τι γίνεται με τον επαναπατρισμό, τι γίνεται με την μετεγκατάσταση και να επιταχυνθεί η αναθεώρηση του Δουβλίνου να μην στιγματίζουν τον κόσμο, να μην τους βάζουμε ταμπέλες, μην στρέφουν τον ένα κατά του άλλου. Ήρθε η ώρα να αλλάξουν το αφήγημά τους οι ηγέτες. Δεν είναι ούτε βάρος, ούτε κίνδυνος. Είναι άνθρωποι οι πρόσφυγες και χρειάζονται προστασία. Ο κύριος Πλέγκοβιτς είναι ο τελευταίος, το Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την επισκόπηση ε, της ε, μεταναστευτικής πολιτικής και ε, του θυματολογίου. Τους τελευταίους μήνες μπήκαν στην Ευρώπη πάνω από 800.000 πρόσφυγες και μετανάστες και φέτος πολλές χιλιάδες ακόμα. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε τώρα ανεξέλεκτες ροές ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από το πόλεμο για να γλιτώσουν τη ζωή τους, αλλά θα πρέπει να το οργανώσουμε αυτό με τρόπο και ανθρώπινο και νόμιμο κυρίως. Γι' αυτό χαίρομαι για τις προτάσεις σας για την αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου για να ε, προστατεύεται η ζώνη Σέγγεν και να ε, ε, γίνεται με τακτικό τρόπο και συγκροτημένο αυτό. Χθες έγινε μια απόπειρα συμφωνίας με την Τουρκία για να προστατεύονται τα σύνορα και θα πρέπει να βοηθηθεί και η Ελλάδα γιατί είναι ικτρή η κατάσταση ε, στα ελληνομακεδονικά σύνορα, λέει ο μιλητής, που θα γίνει και ντόμινο για όλα τα Βαλκάνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω λάβει 17 παρακαλώ αιτήματα για τη διαδικασία Catch the Eye. 17. Δυστυχώς δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους τους συναδέλφους διότι έχουμε καθυστερήσει μεταξύ άλλων και έχουμε και άλλες πέντε συζητήσεις για απόψε. Λοιπόν, με τη σειρά η κυρία Σόιντροβα. Okay. She's not here. Mrs. Virkunen. Λείπει η κυρία Βίρκουνεν θα συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ. Ανησυχώ ιδιαίτερα. Ανησυχώ ιδιαίτερα για την κατάσταση με τη Σέγγεν. Χτες καταλήξαμε σε μια συμφωνία με την Τουρκία, η οποία είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε η Τουρκία θα λύσει τα ευρωπαϊκά προβλήματα με τον μεταναστευτικό. Πρέπει τα εξωτερικά μας σύνορα να προστατευθούν. Έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις, τα hot spot, τα κέντρα υποδοχής, η καταχώρηση, η κατανομή των ε, προσφύγων σε άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε λάβει δεκάδες αποφάσεις και έχουμε υποβάλει δεκάδες συστάσεις, αλλά πού οδηγηθήκαμε σε κράτη-μέλη τα οποία δεν εμπιστεύονται το ένα το άλλο και όπου έχουν ξαναδημιουργήσει ελέγχους στα σύνορα Ακούω τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να εφαρμοστούν με έναν τρόπο που θα βοηθήσουν στο να ξαναλειτουργήσει η Σέγγεν και να μπορεί κανείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κυκλοφορεί ελεύθερα και με ασφάλεια. Αλλά ασφαλή εξωτερικά σύνορα η χώρα μου δείχνει πως η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι ε, λέξεις κενές νοήματος και προσπαθούμε να λύσουμε τη χειρότερη κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι κρίση υπαρξιακή για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είπε σήμερα ο ύπατος αρμοστής ε, για ε, θέματα προσφύγων του ΟΗΕ. Εμείς βοηθάμε την ΕΑΣΟ να επανακαταμείνει τους πρόσφυγες και έχουμε δεχτεί 160 πρόσφυγες από την ε, Ελλάδα παρόλο που ε, συμμάχησαν η Αυστρία και κάποιες χώρες γειτονικέ ε, για να καταστρέψουν τη Σέγγεν και να καταπατήσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευτυχώς η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έδρασε διαφορετικά. Αλλά τι γίνεται με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τι κάνουν η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή και το Συμβούλιο που τιμωρούν την Ελλάδα και την Πορτογαλία γιατί έκαναν, ε, δεν πέτυχαν κάποια δεκαδικά ψηφία στους αριθμούς και δεν κάνουν τίποτα για τα κράτη αυτά τα οποία δεν δείχνουν αλληλεγγύη και επιτρέπουν να βασανίζονται γυναίκες και παιδιά. Γιατί επιτρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκβιάζεται από τον πρόεδρο Ερντοάν. Ευχαριστώ. Ο κ. Κουτσούκ είναι επόμενος ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, κυρία, Πρόεδρο, η Ευρωπαϊκή, κυρία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια κρίσιμη κατάσταση. Είναι πολλά τα κράτη-μέλη που δεν επιθυμούν να μοιραστούν τι ευθύνε και εδώ και μήνε. Έχουμε αναλωθεί σε συζητήσεις για τη συντονισμένη δράση. Παρόλα αυτά δεν ακολουθούμε τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει 700 εκατομμύρια ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια για να δημοσιοποιηθεί το προσφυγικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το σχέδιο δράση με την Τουρκία επίσης έχει το ρόλο του. Είναι απαραίτητο λοιπόν αμέσως να δημιουργήσουμε μια συνοριοφυλακή και μια ακτοφυλακή ε, ευρωπαϊκές και η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα πρέπει να συμμετέχουν για να μην γίνουν απλώς μια ζώνη ασφάλειας ή απομόνωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε μια νέα διαδικασία χωρίς ασύλους στην Ευρώπη. Πρόεδρε, δηλώσεις του κυρίου Τούσκ την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα, τα χρησινά συμπεράσματα του Συμβουλίου και η σημερινή σας ανακοίνωση ε, αποκαλύπτουν ε, την απάνθρωπη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αποσταθεροποίηση, χάος, υπανάπτυξη είναι αυτά που σπήραμε στις χώρες καταγωγής και τώρα θερίζουμε αυτή την κατάσταση. Αυτούς τους ανθρώπους που είναι θύματα. Αυτοί θα απελαθούν ε, χωρίς να είναι ένοχοι, είτε είναι ένοχοι είτε όχι. Αυτή η συμφωνία με την Τουρκία ε, είναι κόλαφος ε, στις διεθνείς συμβάσεις, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις διεθνείς υποχρεώσεις. Και τώρα υποστηρίζουμε και την ατοική πολεμική μηχανή στο Αιγαίο. Οι άνθρωποι αυτοί τι ζητάνε στην Ευρώπη, μια καλύτερη ζωή. το κεφάλαιο ενδιαφέρεται να εκμεταλλεύεται αυτό το φτηνό εργατικό δυναμικό, γι' αυτό τα προκαλεί όλα αυτά. Θα πρέπει να κατανοήσουμε την κρίση και να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Σόλτες, ε, αναφέρατε κύριε Επίτροπε κάποια μέτρα για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης. Επίσης αναφέρατε τη συμφωνία για την επανεκατάσταση ε, μεταναστών και την ανταλλαγή τους με την Τουρκία. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να είναι μια συμφωνία μεταξύ κρατών μελών και θα έπρεπε να είναι το υπαριθμόν ένα μέτρο αυτό, το πρώτο απ' όλα, πριν κλείσουν τα σύνορα και πριν ε, προπάσεις ε, άλλες ενέργειες. Η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών χρειάζεται. Αντί να το κάνουμε αυτό, έχουμε αναθέσει εξωτερικά στην Τουρκία τα θέματα αυτά και είμαστε και πρόθυμοι να πληρώσουμε πολύ υψηλό τίμημα και κυριολεκτικά ε, χρήματα, 6 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Έχουμε κάνει ένα σωρό υποχωρήσει και παραχωρήσει στην Τουρκία σε ό,τι αφορά τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα. Η Τουρκία είναι έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο ε, στη διαπραγμάτευση και στα παζάρια και ξέρει πολύ καλά να τα εκμεταλλεύεται όλα αυτά. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν λοιπόν και να συνοηθούν μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η δεύτερη συζήτηση, λέει ο κύριο Γιούρεκ, για τη μεταμνάστευση που έγινε σήμερα, γιατί ακούσαμε τον φίλο Γκράντη σήμερα το πρωί, που είναι η πατοσαρμοστή. Ε, και παρόλα αυτά, παρόλε τι δύο συζητήσει, ούτε ο ίδιο ούτε ο κύριο Τίμερσον μα ανέφεραν το ποιο είναι το πιο σημαντικό. Πω δεν θα πρέπει να κρύβουμε από τι δικέ μα κοινωνίε πώ έχουν τα πράγματα. Πω η δυναμική ανάπτυξη τη λαθρομετανάστευση στην Ευρώπη έχει φτάσει ρυθμού τη τάξη του 1000% δέκα φορές παραπάνω ε, ελαφρομετανάστες πέταξαν προς την Ευρώπη φέτος και τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν κινδύνους γιατί ακούμε συνέχεια δηλώσεις περί του ανοίγματο ε, νομίμων οδών μετανάστευσης και κάποια οράματα τα οποία τους δημιουργούν την εντύπωση πως έχουν την ευκαιρία. Θα έπρεπε να τους πούμε την αλήθεια. Να μην τους παροτρύνουμε να έρθουν στην Ευρώπη γιατί είναι ανεύθυνο κάτι τέτοιο και θα ήταν αδύνατον για αυτούς που λένε και υπόσχονται τέτοια λόγια να ε, μας εξηγήσουν πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τίμερμανς. Ε, είπατε αν πραγματικά πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να επιλύσει το προσφυγικό πρόβλημα. Είπατε προηγουμένω και κατηγορήσατε την Ελλάδα ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τα σύνορά τη ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος κάθε δίπλα σας και μέχρι πρώτη ήταν υπουργό Άμυνα της χώρας, να σας πει εάν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις δεν είχαν πραγματικά αυτή τη δυνατότητα ή εάν ουδέποτε η ελληνική κυβέρνηση τους ανέθεσε αυτή την αποστολή υπακούοντας σε έξωθεν εντολές μόνο και μόνο για να φτάσουμε σε αυτό το απαράδεκτο σημείο. Μιλάτε για ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή τη στιγμή που η Τουρκία δεν δέχεται να παραλάβει όσους παρανόμως και λαθρέως στέλνει στην Ελλάδα γιατί επιμένετε να εφαρμόσει την αποτυχημένη συνθήκη του δουβλίνου η ελλάδα για να μετατραπεί η όμορφη αυτή χώρα και ο εξαθλιωμένο από τα μνημόνια λαός της σε ένα απέραντο και απαράδεκτο και άθλιο στρατόπεδο συγκεντρώσεως δυστυχισμένων ψυχών; και τέλος γιατί αυτή η αιμονή με την τουρκία η οποία συνεχώς μας εκβιάζει απειλεί και απαιτεί συνεχώς περισσότερες παροχές; κατά την αίσθησή μου το να αναθέσουμε στην τουρκία να προστατεύσει τα σύνορα της ευρώπης είναι σαν να βάζουμε ένα βιαστή να κοιμηθεί με μια γυμνή γυναίκα για να τον βοηθήσουμε να απαλλαγεί από το πρόβλημά του. αν από ιατρική απόψεω αυτό το πείραμα μπορεί να επιτύχει δεν ξέρω. από πολιτική απόψεω όμω σίγουρα όχι. Η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον ε, Επίτροπο για τη σημερινή εισήγηση και για τις καινούργιες νομοθετικές προτάσεις για τις οποίες ε, εγώ σας ε, δηλώνω ότι δεσμεύομαι να κάνω εγώ κάτι για αυτή την ε, κρίση. Οπότε θα πρέπει να τι θα γίνει με τους ε, πρόσφυγες αυτοί που αξίζουν ε, την προστασία. Και έχουμε επίσης και κάποιους κονούς μεταναστές. Δεν μπορούμε να τους καλύψουν, το είπε και την περσμένη εβδομάδα ο κύριος τους και είπε ότι οι οικονομικοί μετανάστες θα πρέπει να μην ταξιδεύουν γιατί δεν είναι δυνατόν να τους φιλοξενήσουμε και δεν μπορούμε ούτε καν να τους υποδεχθούμε. Άρα θα πρέπει να ακολουθήσουν την πραγματική οδό για να επιλύσουμε αυτή την κρίση, κυρίως όσον αφορά το τι γίνεται στη Συρία, αλλά και στη Λιβύη και θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Έτσι ε, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι τρομοκράτες ε, οι οποίοι μαζί με τους μετανάστες χρησιμοποιούν την Βαλκανική οδό. Θα πρέπει μένως να επιστρατεύσουμε όλες αυτές τις εξειδημένες υπηρεσίες, την Europol και την Eurojust. Και έτσι θα πρέπει να προσπαθήσουμε για κάποια ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ τους όλες οι χώρες μέλη, ώστε να φρενάρουν αυτό το φαινόμενο. Και ο τελευταίος είναι ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι πάρα πολλές χιλιάδες Ευρωπαίων αισθάνονται τώρα πάρα πολύ άσχημα γιατί έχουμε ασυνέπεια των αποφάσεων, δεν έχουμε καμία στρατηγική, ε, δεν, έχετε αθετήσει πάρα πολλές υποσχέσεις και δεν δείχνετε καν πολιτική βούληση, δεν δείχνετε καν αλληλεγγύη γιατί το πρόβλημα δεν είναι ούτε οι ποσοστώσεις, ούτε η λύση έγκυται ή στο να συμφωνήσουμε με την Τουρκία και να κάνει η Τουρκία τη διαχείριση προσφύγων και μεταναστών ή επίσης να τάζουμε τον ουρανό μετάστρο. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο. Να πείτε στο Συμβούλιο ότι είναι τερατώδες αυτό το οποίο κάνουν. Να δίνουν υποσχέσεις στην ε, Τουρκία για κάποια πράγματα που δεν μπορούν, ούτε θέλουν να το κάνουν τα κράτη-μέλη. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρόκειται έτσι να εξυπηρετηθούν εάν δεν πιέζονται τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόεδρος. Ο Επίτροπος Αφραμόπουλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εξωτούμε κυρίες και κύριοι. Εν γέννη θα έλεγα ότι συμφωνούμε με κάποιες εξαιρέσεις όλοι ως προς τις βασικές γραμμές για την αντιμετώπιση αυτής της άνευ προηγουμένου κατάστασης. Η χθεσινή συνόδος κορυφής συνιστούσε ένα απαραίτητο βήμα, όχι όμως καταληκτικό καθώς η σύνοδος της προσεχούς εβδομάδας είναι ακόμη πιο σημαντική. Τώρα όλοι ευρίσκονται ενώπιον των ευθυνών τους και όλοι θα κρυθούν και θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Τι πρέπει να επικρατήσει, ποια είναι η κοινή μας αντίληψη εδώ. Μια απτή αλληλεγγύη για όλα αυτά τα θέματα που συζήτησαν εχθέ οι ηγέτε κρατών και κυβερνήσεων. Αλληλεγγύη. Αυτή είναι η βάση, ο κύριο πυλώνα των προτάσεων της Επιτροπής. Η προσφυγική κρίση είναι καταλήτης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα σας υπενθυμίσω εδώ το μύθο του Σισίφου, που όλοι γνωρίζετε. Γίνεται την Ευρώπη τώρα στη θέση του Σισίφου. Ναι, η Ευρώπη κουβαλάει ένα μεγάλο βάρος στους ώμους της. Είναι απαραίτητο όμως όλα τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν την Ευρώπη να ανεβάσει αυτό το αγκονάρι στην κορφή. Να μην την αφήσουν να το εγκαταλείψει και να κυλήσει πίσω στην πλαγιά. Να μην γυρίσει πίσω. Η τάση για μια εύκολη λαϊκιστική ρητορία φαίνεται σε όλες τις χώρες που είχαν εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο μόνο ο εξτρεμισμός, ο εθνικισμός και η ξενοφοβία μπορούν να κερδίσουν έδαφος εις βάρος των ιδεωδών και των αξιών της Ευρώπης. Θα επαναλάβω, δεν πρόκειται να αλλάξουμε στρατηγική και καλούμε τους πάντες να την τηρήσουν. Χρειαζόμαστε μεγάλης κλίμακας επανεκαταστάσεις, ουσιαστική, πραγματική επαναπροώθηση όσων δεν έχουν δικαίωμα προστασίας, ισχυρά εξωτερικά σύνορα και σε αυτό όλα τα κράτη-μέλη συμμερίζονται τις ίδιες ευθύνες. Την ευθύνη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τη διαφύλιση του Σέγγεν. Και αν δεν αναγνωρίζουν κάποιοι τη συμβολική αλλά και πολιτική αξία του Σέγγεν κάποια κράτη και τις δικές τους ευθύνες, θα πρέπει μη τι άλλο να αναγνωρίσουν το οικονομικό κόστος της απουσίας του Σέγγεν. Δεν θα επαναλάβω τις ε, απόψεις μου και τις ιδέες μου για το Σέγγεν, τις γνωρίζετε όλοι η μεταναστευτική πίεση είναι τέτοια κλίμακα που κανένα κράτο μέλο μόνο του δεν θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Χρειαζόμαστε αμέση υποστήριξη προ όλε τι επιχειρήσει τη Frontex και ταχύτατη συμφωνία για μια, ε, πρόταση για τι ακτοφυλακέ και τι συνοριοφυλακέ τη Ευρώπη. Κανεί δεν μπορεί μόνο του να τα καταφέρει καλύτερα και αν δεν συμφωνήσουμε, αν δεν στρατευθούμε όλοι, δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Και σε αυτό έρχεται και η στράτευση και προσήλωση των εταίρων μας. Τη είπα της Αρμοστίας των ΗΠΑ για τους ε, πρόσφυγες του ΝΑΤΟ, το οποίο θα σταματήσει τις δραστηριότητες των λαθροδιακινητών. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κηρύξει πόλεμο κατά των λαθροδιακινητών. Και βέβαια των κρατών που έχουν θέσει κλειδί όπως η Τουρκία. Ναι, βεβαίω, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια τη Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε αυτή την παγκόσμια κρίση. Ξέρω ότι ορισμένοι μπορεί να έχουν ε, επιφυλάξεις ή και αμφιβολίες. Παρ' όλα αυτά είναι παίκτη με θέση κλειδιού η Τουρκία σε όλη αυτή την υπόθεση και αμφιβολιες παρολα αυτα ειναι παικτη με Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δράσουμε όμω αντίθετα με του κανόνε μα και αυτό θα καταστεί σαφέ κατά τι προσεχεί ημέρε που θα οδηγήσουν προ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η επαναπροώθηση μπορεί να γίνεται μόνο με απόλυτη συμμόρφωση στο διεθνέ δίκαιο και το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη στρατηγική μας. Η επανεκατάσταση είναι μια, η πρώτη μας, η κυρία μας προτεραιότητα και όπως είπα και στην ακρόασή μου πρέπει να οικοδομήσουμε νόμιμους τρόπους για όσους έχουν ανάγκη να φτάσουμε μέχρι την Ευρώπη. Το ταχύτερο δυνατό όπως υποσχεθήκαμε θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και συμφωνώ μαζί σας ότι χρειάζεται ένα ισοδίκαιο σύστημα επιμερισμού των βαρών και τη νόμιμη μετανάστευση. σε έναν κόσμο μεγάλης κινητικότητας δεν μπορούμε ε, να έχουμε μια Ευρωπαϊκή ε, Ένωση χωρίς μια ε, πραγματική πολιτική για την μετανάστευση και τη διεθνή συνεργασία βέβαια. Και βέβαια η συνεργασία και με τρίτες χώρες, ο συντονισμός με τον οικονομικό τομέα. Και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό περισσότερο συντονισμένη πολιτική για την κοινωνική ενσωμάτωση που θα συμπληρώσει αυτή την εικόνα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι τοποθετήσεις μου ήταν πολύ χρήσιμες. Σας ευχαριστώ. Και ως φίλο της λαμβάνω σοβαρότατα υπόψη εν των προσεχών εξέλιξεων. Εδώ μέσα στο σώμα γεννήθηκε αυτή η πολιτική μας. Εδώ μέσα στο κοινοβούλιο θα προστατέψουμε και θα υπερμηνθούμε αυτή τη πολιτική στο όνομα των ευρωπαϊκών αξιών, στο όνομα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ε, στη... Θα πρέπει να συζητήσουμε, μάλλον, σε σχέση με τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών